Kolleginnen und Kollegen, ich heiße alle ganz herzlich willkommen. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτούς που κατάφεραν να έρθουν Βεβαίω δεν είναι ότι έχουμε υπερβολικά πολύ κόσμο ακόμη εδώ, αλλά αρκετοί είναι ήδη εδώ. Σήμερα έχουμε ακρόαση, όπως ξέρετε, Σήμερα η συνεδρίασή μας αυτή, η ακρόαση, ε, δεν μαγνητοφωνείται αλλά περνάει στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το περίφημο web streaming που λένε. Ε, στο τέλος των εργασιών μας θα μπορέσουμε να πιούμε ένα κοκτέιλ εδώ έξω από την αίθουσα είναι η πρώτη μέρα του hearing βεβαίω σήμερα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εμπειρογνώμονες που βρίσκον, που βοήθησαν μέχρι τώρα, αλλά βρίσκονται και που, βρίσκονται σήμερα και εδώ. Ε, τώρα εδώ βλέπετε το πρώτο πάνελ, αύριο θα υπάρχουν άλλα δύο πάνελ, τρία είναι συνολικά. Nicht mehr, um, viel Δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, φαντάζομαι, για την εντολή της ειδική Επιτροπής SURE, της Επιτροπής μας. Το δι... Η ομολομέλεια μας έδωσε διάφορες εντολές να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες και να εφαρμόσουμε προτεραιότητες νομοθετικής και ε, από νομοθετική αλλά και ουσιαστική άποψη πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε πια. Ε, οι κρήματοδοτικά ε, εργαλεία είναι απαραίτητα, πια δεν είναι, να χαράξουμε κατευθυντήριες γρομ κατευθυντήριες γραμμές, να χωρίσουμε τα πράγματα σε κατηγορίες ανάλογα με τη σημασία του ή με το θέμα τους και να σκεφτούμε να το θέμα των εσόδων ιδιαίτερα για να απαντήσουμε στο τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής μας το πολύ βασικό ερώτημα χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση ή όχι. Τώρα είπα στο τέλος της συνεδρίασης, το τέλος θα είναι η Ολομέλεια του Ιουνίου. Το τέλος λοιπόν θα πρέπει να έχουμε καταλήξει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις με την MFF έναντι του Συμβουλίου ναι, και θέλουμε να έχουμε μία θέση αλλά να έχουμε διεξάγει και συζητήσεις τέτοιες τους ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι λέμε ότι δουλεύουμε παράλληλα με το Συμβούλιο αλλά η παραλληλία δεν είναι αυτή που είναι στη γεωμετρία που οι παράλληλες δεν συναντώνται ποτέ θα θέλαμε κατά τη διάρκεια των εργασιών να συναντιόμαστε με το Συμβούλιο να ανταλλάσσουμε απόψει. και με την Επιτροπή υπάρχει, ξέρετε, για τη Task Force που έχει δημιουργηθεί για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και βεβαίως δεν πρόκειται να επανεφεύρουμε τον τροχό. Ήδη έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και ξεκινάμε βασιζόμενοι σε μια πολιτική που τουλάχιστον επί χάρτου υφίσταται και δει με πολύ ευρεία ευρωπαϊκή συνένεση και που Κάποιοι την ονομάζουν στρατηγική 2020. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει πάρει τις αποφάσεις του. Εμείς ε, ε, γνωμοδοτήσαμε και δει θετικά υπέρ της απόφασης αυτής η Ευρώπη του 2020, η έξυπνη ανάπτυξη, η ε, καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη, η οικολογική Ευρώπη, η προώθηση της ε, οικονομίας όμως με κοινωνικό πρόσωπο, με θέσεις εργασίας κτλ. Όλα αυτά, οι, όλοι αυτοί οι στόχοι είναι οι στόχοι στρατηγικής του 2020 που υποδιαιρούνται σε τρεις ομάδες, αν θέλετε, θεματικές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευθούν. Τα έχουμε συζητήσει αυτά στο παρελθόν. Τα συζητήσαμε και στη Ρήγα και είπαμε ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν σωστά όχι μόνο αν καθίσουμε και σκεφτούμε όλους τους στόχους μαζί α, ο, αλλά και αν καταφέρουμε να συνεργαστούν όλα τα επίπεδα μαζί και όταν υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των ενδιαφερόμενων των προσπαθειών και τα λοιπά. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Πρέπει αν καθίσουμε να σκεφτούμε ποιες δυνατότητες έχουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας ε, θα δούμε ότι τα κύρια εργαλεία μας είναι τρία, συντονισμός, ε, συνεργασία και προϋπολογισμός. Και ο ε, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άποψή μου παίζει ρόλο κλειδί στην εφαρμογή της στρατηγικής μας και στην επίτευξη των στόχων. Η στρατηγική αυτή Βεβαίω και το κατά πόσο θα επιτευθούν οι στόχοι της στρατηγικής αυτής θα είναι ε, βεβαίως και η βάση για την περαιτέρω πορεία μας. Ξέρουμε όλοι ότι οι δαπάνες ε, είναι μοναχά 2% στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Μιλάμε για δημόσιες δαπάνες, ε? όμως πιστεύουμε ότι παρόλο που δεν είναι μεγάλο ποσοστό του προπολογισμού πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει καλύτερη συνεργία μεταξύ των δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Οι επενδύσεις βεβαίως μέσα στα πλαίσια της Αττικής 2020 θα πρέπει να προέλθουν από στο, από το εθνικό επίπεδο προφανώς αλλά παρακολουθούμε κι εμείς ο μικρός προϋπολογισμός λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μικρός πράγματι παρόλο που σε απόλυτε τιμές μπορεί να φαίνεται μεγάλος ο μικρός λοιπόν προπολογισμό μας πρέπει να οδηγήσει στη μεγαλύτερη δυνατή πρόσθετη αξία και πρέπει να βοηθήσει επίσης το να επιτευχθούν οι στόχοι. Βέβαια η οριστική μορφή της στρατηγικής 2020, Ευρώπη 2020 δεν ε, ε, έχει ε, αποφασιστεί ακόμη, βρισκόμαστε στο στάδιο των συζητήσεων κτλ. Αλλά ένα είναι σίγουρο ότι όλες οι κοινοτικέ πολιτικές και η αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής και η εξωτερική πολιτική, όλες οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν τη στρατηγική του 2020. Και υποθέτω ότι όλοι εδώ συμφωνούμε ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι η στρατηγική πολιτική για την επόμενη δεκαετία. Και είναι και το σημείο αναφοράς μας βεβαίως και για τις ε, προοπτικές, ε, δημοσιονομικές προοπτικές τα λοιπά. έχουμε συζητήσει αυτά. Ich Υπάρχουν βεβαίως από εκεί και πέρα και άλλα εργαλεία όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, η αγροτική πολιτική, το πλαίσιο, το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα κτλ. Α, εργαλεία τα οποία και αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε και να τα αλλάξουμε ενδεχομένως για να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματά τους. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, θέλουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, θέλουμε να δημιουργήσουμε, επαναλαμβάνω, την πρόσθετη αξία, την υπεραξία που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Ζητώ από τους εμπειρογνώμονες που βρίσκονται μεταξύ μας να αρχίσουν να σκέφτονται λίγο με κριτικό πνεύμα με έναν διαφορετικό εφάνταστο τρόπο γιατί μας ενδιαφέρουν και οι επικρίσεις και με κυρίως οι καινούργιες ιδέες για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Ποιες δραστηριότητες μπορεί, πρέπει να εγγραφούν στον προπολογισμό, ποιες δεν χρειάζεται να εγγραφούν, να δεσμευτικά αν θέλετε στο προπολογισμό και μπορούν να προωθηθούν από τα κράτη-μέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη τελευταία ανάλυση εδώ πρόκειται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Και βεβαίως δεν μπορούμε να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε το μέλλον της Ευρώπης όταν ξέρουμε ότι υπάρχει το 2014 όπου κάποια πράγματα θα αλλάξουν. Έτσι. Γι' αυτό η στρατηγική Ευρώπη 2020 ουσιαστικά είναι μια στρατηγική που μας αναγκάζει ήδη από τώρα να φτιάξουμε ένα μοντέλο ε, που θα εφαρμοστεί στο μέλλον, όχι άμεσα, ένα μοντέλο οικονομίας της αγοράς με κοινωνικό πρόσωπο. Αυτά, σαν εισαγωγή. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας. Θα υπάρχει κάποιος που θα διευθύνει τη συζήτηση, ο moderator, ο οποίος θα δίνει το λόγο και θα σας και θα ζητεί απαντήσεις και αναπάνελ θα έχουμε τρεις με τέσσερις εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα να πω όμως ε, πρώτα-πρώτα μερικά πρακτικά οργανωτικά πράγματα. Πώς φανταζόμαστε την ακρόαση. Κατά τη διάρκεια του πάνελ, ο moderator θα κάνει μια εισαγωγή 5 λεπτά και μέσα αυτό 5 πεντάλεπτο θα θέτει τα ερωτήματα τα οποία θα ήθελαν να απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες. Και μετά οι εμπειρογνώμονες, ο κάθε εμπειρογνώμονας θα έχει 5 λεπτά καιρό να απαντήσει στα ερωτήματα. και μετά οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές ε, θα θέσουν τα δικά τους ερωτήματα. Θα θέλαμε να γίνει ζωντανή συζήτηση. Δεν θα θέλαμε να γίνουν απλώς δηλώσεις ή ομιλίες από τους ευρωβουλευτές αλλά να τεθούν ερωτήματα για να απαντηθούν και να ξανατεθούν ερωτήματα κτλ. Ο... Τα ερωτήματα των ευρωβουλευτών ε, πρέπει να τίθεται μέσα σε δύο λεπτά. Βεβαίως ο moderator θα οργανώσει την περαιτέρω ροή των συζητήσεων. Θα δούμε βεβαίως τι θα γίνει με το χρόνο. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται δεύτερος και τρί... δεν θα χρειάζεται δεύτερος και τρίτος γύρος από πλευράς αυλοβουλευτών και δεν ε, νομίζω ότι θα πρέπει να τεθούν μοναχά να τεθεί μοναχά μία ερώτηση από του, τους παρεμβαίνοντες ή τις παρεμβαίνουσες θα μπορούσε κανείς να θέσει και δεύτερη, δεύτερη και τρίτη ερώτηση. Αυτά για το πώς φανταζόμαστε την πρακτική οργάνωση. Τώρα, ξεκινάμε με το πρώτο πάνελ. Χαιρετίζω εδώ τον καθηγητή Αντρέζα Πύρ, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνούς οικονομίας και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Καλωσορίζω τον κύριο Πατρίκ Πρέσλερ, ο οποίος είναι διευθυντής της ε, Fraunhofer Gesellschaft εδώ στις Βρυξέλλες, τον κύριο Χωσέ Ράις, που είναι διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Κοίμπρα στην Πορτογαλία και χαιρετίζω και τη μόνη γυναίκα σε αυτό το πάνελ, την κυρία Λέσλι Βίλσον, που είναι η Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων και τον ε, moderator, τον Ανδρέα Ρέντα, ο οποίος προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικών Σπουδών. Η σειρά σα τώρα κύριε Ρέντα. Thank ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επίσης για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε σε αυτό το ενδιαφέρον πάνελ και μάλιστα να διευθύνω για τη συζήτηση κάτι το οποίο θα είναι εύκολο και ενδιαφέρον λόγω της ικανότητας και της δυνότητας των συμμετεχόντων. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Ροντρίγκε που μου ζήτησε πρώτος να έρθω εδώ. Ο τίτλος του πάνελ αναφέρεται στην έξυπνη ανάπτυξη. Τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις λέξεις έξυπνη, αηφόρα, και ε, την φράση «μη αποκλεισμό στην οικονομία και στην ανάπτυξή της. Περνάμε από μια δεκαετία η οποία είχε σαν στόχο την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πιο καινοτόμο και τεχνολογικά προηγμένη κοινωνία, βασισμένη στη γνώση. Προφήσαμε και σε αυτή τη δεκαετία την ιδέα της αηφορίας και όλους αυτούς τους στόχους τους δώσαμε διαφορετικό βάρος κατά περίπτωση βέβαια, ανά περίοδο χρονική θα έλεγα, αλλά χαρακτήριζαν συστηματικά τον πυρήνα της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Σήμερα έχουμε μια νέα ατζέντα, μια νέα στρατηγική, τη στρατηγική 2020. Είναι μια πολύ φιλόδοξη στρατηγική αν δει κανεί ποιε είναι οι βασικές πρωτοβουλίε αυτή της στρατηγικής, μία από αυτές, η ψηφιακή, ε, θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή οικονομία η οποία ξεπερνά το πρόγραμμα που οδήγησε στην Ευρώπη ε, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς από το 1992 και μετά. Τεράστια σημασία λοιπόν, προσπαθούμε εδώ και χρόνια να κλείσουμε βέβαια το θέμα της εσωτερικής αγοράς, και έχει φτάσει η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτή η συζήτηση, γιατί οι συζητήσεις μέχρι τώρα για την αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών προοπτικών θα ξεκινήσουν σε λίγα χρόνια, από το 2014 και μετά, αλλά το μέλλον είναι εδώ. Η κατανομή των προϋπολογισμών και οι πρωτοβουλίες διακυβέρνησης θα αποφασιστούν τώρα που ξεκινάει η στρατηγική του 2020 και αυτό θα καθορίσει την επιτυχία ή μη της στρατηγικής αυτής. Η πρώτη ερώτηση είναι αν μπορεί η Ευρώπη να χάσει για μια ακόμη φορά τους στόχους που θέτει. Όταν μιλάμε για τον καθορισμό των πολιτικών λέμε ότι ό,τι προσμετράται ολοκληρώνεται. Αυτό έχει συμβεί τις προηγούμενες δεκαετίες όταν εκπληρώσαμε κάποιους από τους στόχους τους οποίους είχαμε καθορίσει στα πλαίσια της ατζέντα της Λισαβόνας. Στον τομέα της γνώσης και της καινοτομίας υπήρξαν προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα αυτά τα οποία αναδύθηκαν και στα πλαίσια της πρότασης για τη Λισαβόνα και στα πλαίσια της ευρύτερης πρότασης ε, που φάνηκαν τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι ότι δεν είναι απαραίτητα ένα πρόβλημα μεγέθους του προϋπολογισμού σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Πολλοί σχολιαστές είπαν ότι σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης στην έρευνα και ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πίσω από άλλες χώρες οι οποίες είναι ηγέτιδες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας όπως είπα. Και η ιδιωτική πλευρά είναι αυτή η οποία θα πρέπει να δώσει περισσότερα κίνητρα. Είδα στους υπολογισμούς για τη στρατηγική 2020 ότι μία αλλαγή τα επόμενα χρόνια πάνω στην οποία θα βασίσουμε ε, την ευρωπαϊκή οικονομία είναι τα venture capitals. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σε επίπεδο δημόσιων δαπανών έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα σωστό σύστημα συνεργασίας με τα venture capitals και ταυτόχρονα έχουν δημιουργηθεί και νέα προβλήματα στην λεγόμενη διαχείριση της καινοτομίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί γιατί το θέμα της χρήσης του δημόσιου χρήματος στον τομέα της καινοτομίας δεν πρέπει να παραμείνει στο ίδιο στάδιο που βρίσκεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προβλήματα της διακυβέρνησης ήταν και οριζόντια στις Βρυξέλλες ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα χρήματα οι Βρυξέλλες και πολυεπίπεδα, οι σχέσεις δηλαδή ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη-μέλη μεμονωμένα. Υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα σε σχέση με την υπερβολική κατανομή πολλών προγραμμάτων και πολλών κεφαλαίων δημιούργησε μία πολυδιάσπαση σε σχέση με το δημόσιο χρήμα ε, που είχε σαν στόχο την γνώση και την ανταγωνιστικότητα. Αυτή η πολυδιάσπαση θα πρέπει να αποφευθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτή η αποσπασματοποίηση και ένα άλλο σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε καλοί στην ανάπτυξη της γνώσης, αλλά δεν μπορούμε να μετατρέψουμε την γνώση σε καινοτομία. Κάνουμε κάτι στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 για να βοηθήσουμε τη μετατροπή της γνώσης στην καινοτομία και την εμπορία νέων προϊόντων άραγε. Και αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι ομιλητές μας. Ταυτόχρονα υπήρξαν διαφορετικά προβλήματα στο παρελθόν, στα πλαίσια των μικρομεσαίων, που είναι ο πραγματικός κινητήρας της αλλαγής στην ευρωπαϊκή κοινοτομία. Εγώ ηγούμενος σε μία σειρά στροκύλων τραπεζών για τις μικρομεσαίες άκουσα ότι τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να αντιμετωπίζουν ένα διαφθορτικό πρόβλημα γιατί το μικρότερο πρόγραμμα το οποίο μπορούν να καλύψουν είναι πολύ μεγάλο για να καλύψει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό διορθώνεται με τις νέες προτάσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε για να συμπεριλάβουμε τις μικρομεσαίες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε πόσο συντονισμένη θα πρέπει να είναι η δαπάνη και πόσο μπορεί ο συντονισμός αυτός να είναι αποδοτικός. Να δούμε επίσης και πόσο ε, δαπανώνται τα χρήματα στα κράτη-μέλη και στα διαφορετικά ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για τη βελτίωση της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των μεγάλων προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν σημασία για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της ε, ε, καινοτομίας ε, και της γνώσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τμήματα και της δικής σας συζήτησης. Υπάρχει μια κάποια βεβαιότητα σήμερα σε σχέση πόσο ε, συγκεντρωτική ή πόσο αποσπασματική θα πρέπει να είναι η διαχείριση της πολιτικής αυτής. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να διακυβερνώνται με συγκεντρωτικό τρόπο ή θα πρέπει να υπάρχουν μεμονωμένες στρατηγικές οι οποίες να ορίζουν τη διαχείρισή τους. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτές τις κύριες μορφές χρηματοδότησης, πώς αυτές οι επτά πρωτοβουλίες να μπορέσουν να ανθίσουν και να γίνουν αντικείμενο ε, καλής διαχείρισης έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει τους στόχους της. Σε αυτή τη φάση δεν θα πω περισσότερα οι συμμετέχοντες στην τράπεζα θα μπορέσουν να εκφράσουν τις θέσεις τους ελεύθερα. Αυτό που μπορώ να αποκλίνοντα την εισαγωγή είναι ότι είδα αρκετές ερωτήσεις οι οποίες διανέμονται από τους οργανητές που απευθύνονται στους συμμετέχοντες στο πάνελ. Η πρώτη που μου έκανε εντύπωση ήταν μια εξαιρετική ερώτηση. Αν είχατε ένα δις ευρώ και είχατε τη δυνατότητα πώς να δαπανίσετε, πού να βάλετε τα χρήματα αυτά για να βελτιώσετε τη γνώση και την καινοτομία στην Ένωση. Τι θα κάνατε, προς ποια κατεύθυνση. Θα δούμε τι ιδέες έχουν οι πανελίστες. Δεν μιλάμε για ένα δις εδώ, μιλάμε για πολύ περισσότερα χρήματα και για τις πιθανές επιρροές τους στην ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι τιμή λοιπόν τώρα για μένα να δώσω αμέσως το λόγο στον καθηγητή Αντρέ Σαπίρ για την εισαγωγική πεντάλεπτη παρουσίασή του. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Πρόεδρο για την ευγενή πρόσκληση που μας απίφθηνε να είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα. Στο τέλος της σύντομης παρουσίασής μου θα απαντήσω το ερώτημα για τον εκατομμυριούχο ή τον πολύ εκατομμυριούχο, αλλά τέλο πάντων. Αντρέα, θέλω να πω ότι μόλι ανέφερε ότι έχουμε μια στρατηγική δεκαετίας που δεν πέτυχε τα αποτελέσματά της. Μιλώ για τη στρατηγική της Λισαβόνα. Έχουμε τώρα μπροστά μας μια νέα στρατηγική δεκαετούς επίσης ε, ορίζοντα. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι φυσικά και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να περιμένουμε μία ακόμα δεκαετία για να δηλώσουμε ότι δεν πετύχαμε με τη νέα στρατηγική. Διότι ταυτόχρονα προχωρούμε και προχωρούμε πολύ αργά θα έλεγα, ενώ άλλοι κινούνται πολύ πιο γρήγορα. Εμείς πάμε σαν τα σαλιγκάρια και άλλοι τρέχουν. Αυτό που μπορούμε λοιπόν ε, να, πούμε είναι ότι η κρίση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε διχασμό, ε, σε διχοτόμηση στις κοινωνίες. Αυτό το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη είναι και φύση ανάπτυξη αλλά και ανάπτυξη εν γέννη. Χωρίς ανάπτυξη δεν θα λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη και ούτε βέβαια θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, για τη θέση που θέλουμε να έχει η Ευρώπη σε αυτή την ταχύως μεταβαλλόμενη οικονομία, χωρίς καινοτομία και ευφύ ανάπτυξη προσανατολισμένη στην καινοτομία. Άρα η άποψή μου είναι ναι, βεβαίως ε, και είμαστε υπέρ στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, αλλά πρέπει να είναι αξιόπιστη η στρατηγική αυτή και δεν θα πρέπει να κάνουμε λάθος. Διότι και ο ιδιωτικός τομέας αμφιβάλλει τα μάλλα για το κατά πόσον ε, ε, η στρατηγική αυτή η, δεκαετού, η δεκαετής είναι αξιόπιστη περισσότερο ή το ίδιο με την προηγούμενη. Και όπως είπα, είμαι υπέρ της στρατηγικής αυτής, αλλά είμαι υπέρ μόνο εάν φέρει αποτελέσματα, εάν είναι αξιόπιστη. Πώς λοιπόν μπορούμε να χαράξουμε μια αξιόπιστη πολιτική, στρατηγική μάλλον, όχι με ωραία λόγια. Να μιλήσουμε για την καινοτομία στην Ευρώπη, ωραία είναι αυτά. Αλλά αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις, δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα απτό. Και πάλι δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ευρώπη στον τομέα αυτό πρέπει να δρά μόνο ή κυρίως μέσω του προπολογισμού της. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι δράσης που θα είναι κυρίως ρυθμιστικό χαρακτήρα. Πού όμως θα κριθεί κάποιος, πού θα δει κάποιος, πού λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις, σκληρές ενδεχομένως, στον προπολογισμό. Όλα τα άλλα είναι φροφρού και αρώματα. Και εκεί, στον προπολογισμό, φαίνονται οι κατευθύνσει που παίρνει κάποιο. Η δική σα λοιπόν ευθύνη είναι τεράστια. Μιλώντας λοιπόν για προπολογισμό, μιλώντας ε, για χρήματα, γνωρίζουμε ότι δεν είναι μεγάλος ε, ο ευρωπαϊκός προπολογισμός, ούτε από ό,τι φαίνεται θα αυξηθεί σημαντικά. Δεν είναι όμως ε, συμβολικός απλά, να πούμε δηλαδή ότι είναι το 2,5% των συνολικών δαπανών σε επίπεδο Ευρώπης, άρα είναι συμβολικός. Όχι. Είναι η εικόνα που θέλει να δώσει για τον εαυτό της η Ευρώπη. Τι θέλουμε να κάνουμε από κοινού, ποιο είναι το όραμά μας, ποιο είναι το σχέδιό μας. Και πέραν αυτού βέβαια είναι σαφές ότι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός θα πρέπει να δράσει ως ένας μοχλός σίγουρα ε, στην κοινοτομία, στην έρευνα. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα κονδύλια δαπανώνται είτε σε εθνικό είτε ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο. Ακόμη και αν δηλαδή ο ευρωπαϊκό προβολισμό δεκαπλασιαζόταν, ήταν το 10% ας πούμε των δαπανών της Ευρώπης πάλι θα ήταν μόνο 10%. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ένας μοχλός, ως διευκολυντής πρέπει να δρά και κατά την άποψή μου δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσουμε να ευθυγραμμίσουμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς στον ευρωπαϊκό. Αυτό θα έρθει από μόνο του. Η Ευρώπη δίνει τις κατευθύνσεις. Τα κράτη-μέλη πιστεύω ότι θα επιδείξουν αρκετή ευφυΐα για να ακολουθήσουν την πορεία την οποία εμείς χαράζουμε από κοινού. Τρίτο σημείο στα πέντε που έχω να αναφέρω. Έρευνα και καινοτομία και τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Βλέποντας την Ευρώπη, βλέπω ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό ατού, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, που είναι η ενιαία μας αγορά, το μέγεθος της αγοράς μας, το μέγεθος του πληθυσμού μας, η ποιότητα της εκπαίδευσης του πληθυσμού μας εν γέννη. Έχουμε 27 χώρες μέλη, τεράστια ε, πολυμορφία, διαφοροποίηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν μιλά κανείς για καινοτομία και έρευνα. 27 χώρες, 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Συνήθως με καλή εκπαίδευση. Και αυτό πραγματικά είναι μια τεράστια δεξαμενή ταλέντων για την έρευνα και την καινοτομία και για το καθήκον που έχουμε να φέρουμε σε πέρας. Δηλαδή, ότι το πλεονέκτημα αυτό που έχουμε πραγματικά μετατρέπεται σε δυνατότητα, σε δυναμικό. Και αν να δώσει και αποτελέσματα στην έρευνα και στην καινοτομία. Πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν το πλαίσιο, οι συνθήκε πλαισίου. Και παραλαμβάνω, η έννοια αγορά και ό,τι κινείται γύρω από αυτήν και η κινητικότητα δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και πάλι όμω εδώ μπορεί να βοηθήσει ο προπολογισμό. μπορούμε να ελπίσουμε θα βοηθήσει. Εάν μιλάμε λοιπόν για έρευνα και καινοτομία, κατά την άποψή μου υπάρχει μία λέξη κλειδί. Αριστεία. Δεν μπορεί να υπάρχει έρευνα και καινοτομία χωρίς να δοθεί έμφαση στην αριστεία. Στον ανταγωνισμό δηλαδή. Καταλαβαίνω ε, ότι θα υπάρξει άμεσα ε, κάποια κριτική σε αυτά που λέω, είτε από κάποιους από εσάς, είτε και από κάποια κράτη-μέλη. Δηλαδή θα πει κάποιος ότι άπαξ και αρχίσουμε να αναθέτουμε, να κατανέμουμε τα κονδύλια με βάση τον ανταγωνισμό και την αριστεία, ίσως ε, αυτή η κατανομή, αυτός ο επιμερισμός να μην είναι ισομερής σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάποιος θα πει μήπως αυτό είναι άδικο. Αυτό που έχω να απαντήσω στο ερώτημα αυτό είναι ότι αυτή η ατζέντα, η ατζέντα του 2020, κάνει λόγο για ευφύ ανάπτυξη, αλλά και για βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη για όλους. Ναι, φυσικά και έχουμε στόχους. Δεν είναι η ευφύς ανάπτυξη ο μόνος στόχος, έχουμε και άλλους στόχους. Βιωσιμότητα, η συνοχή, αλληλεγγύη. Έτσι πρέπει να είναι. Αλλά για τα εργαλεία τα οποία είναι προσανατολισμένα στην έρευνα και την καινοτομία, εκεί θα πρέπει οι πόροι να διατεθούν προς την αριστεία, με γνώμονα την αριστεία. Γνωρίζοντας, επαναλαμβάνω, ότι έχουμε αυτό το δυνάμει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Επιμένω λοιπόν στην ανάγκη να τονίσουμε την σημασία της αριστείας. Να δώσουμε λοιπόν έμφαση κατά συνέπεια και στον ανταγωνισμό που είναι χέρι με χέρι με την αριστεία. Και έρχομαι τώρα στο πέμπτο σημείο και να απαντήσω ε, στο ερώτημά σας. Αν είχα ένα δισεκατομμύριο ευρώ, πού θα τα επένδυα, πού θα τα έβαζα. Σε μια μελέτη που κάναμε με κάποιους συναδέλφους για τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, ακριβώς κάναμε την πρόταση του ενός δεκατομμυρίου ευρώ στο τέλος ε, του εγγράφου μας. Ε, και η πρότασή μας ήταν η εξή. Σε όλα τα συστήματα, τα εκπαιδευτικά μπορούμε την διδασκαλία να τη συνδέσουμε σε έρευνα. Πού μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι στα σχολεία. Αυτό λείπει στην Ευρώπη. Όταν πρέπει λοιπόν να διατεθούν πόροι ανταγωνιστικά σε κάποια προγράμματα εκπαιδευτικά, λέμε ας βάλουμε σε καθένα ένα εκατομμύριο ευρώ. Οπότε θα έχουμε χίλια προπτυχιακά προγράμματα. Και φτάνουμε στο ένα δισεκατομμύριο έτσι. Είπαμε, υπάρχουν, αν δει κανεί, περίπου 50 τομείς έρευνας. Ας επιλέξουμε με επιλεκτική διαδικασία, διαδικασία ανταγωνιστική. Ας επιλέξουμε 20 τμήματα στην Ευρώπη, σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Βέβαια έτσι ξέρουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε πολλά πανεπιστήμια και πολλά προγράμματα. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ λοιπόν για αριστεία μέσω προπτυχιακών προγραμμάτων. Ένα εκατομμύριο ευρώ σε χίλια τμήματα ανά το Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέ. Πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Λοιπόν, Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν ερωτήσεις πολλές από το ακροατήριο. Προχωρώ τον επόμενο μιλητή, Αν θέλετε κι εσείς να απαντήσετε, ευχαριστώ. Το ερώτημά μου ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ. Και κάπου νιώθω λίγο άσχημα γιατί μιλώ μετά τον καθηγητή Σαπίρ, ο οποίος είπε σχεδόν όλα αυτά που είχα ετοιμαστεί να πω κι εγώ. Όταν με προ πρωτοπήρα την πρόσκλησή σας και κοίταξα περί τίνος πρόκειται. Αναφέρεται βεβαίως... Ε, σκέφτηκα ότι ναι, πρέπει να δούμε τι έγινε στο παρελθόν για να μπορέσουμε να κάνουμε το άλμα προς το μέλλον. Ε, πραγματικά η αριστεία και η καινοτομία βασίζεται στον ανταγωνισμό. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό αξίωμα αν θέλετε. Σε μια λοιπόν κατακαιρματισμένη αγορά ε, δεν μπορούν να επιτευχθούν τα πράγματα αυτά. Η αριστεία επιτυχάνεται με συνεργασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όντως μια περιοχή ανεπτυγμένων χωρών που συνεργάζονται και που θα πρέπει να συνεχίζουν να συνεργάζονται. Στο τελευταίο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα ε, αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και αναφέρεται και εκεί η έννοια της αριστείας η οποία... Αλλά Κοιτάξτε, η πρωτοπόρα έρευνα δεν είναι μοναχά θεμελιώδης βασική έρευνα, αλλά κατά κύριο λόγο εφαρμοσμένη έρευνα και σε τομείς ε, μηχανικής. Ε, βρισκόμαστε στην Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν λοιπόν έχουμε ακούσει ε, για το ευρωπαϊκό παράδοξο όπου υπάρχει αριστεία, υπάρχει αρκετά υψηλή χρηματοδότηση που όμως διατίθεται στη βασική έρευνα αλλά νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα, ε, διείσδυση σε νέες αγορές κτλ. δεν βλέπουμε. Τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά εκεί αποτελέσματα έρευνας μπορεί να υπάρχουν στην Ευρώπη αλλά ε, δεν ξέρουμε εάν ε, δεν ε, καταλήγουν στην αγορά στην Ευρώπη όπως καταλήγουν σε άλλες χώρες στην Ασία και στην Αμερική η επίπεδη οθόνη είναι ένα καλό πράδειγμα εδώ η, τώρα για να δούμε την έρευνα η βασική έρευνα θεμελιώδης έρευνα είναι πολιτικά ασφαλής. Γίνεται αποδεκτή από το κοινό δέχονται ότι πραγματικά πρέπει να γίνει βασική έρευνα γιατί αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες εφαρμογές. Αυτό το μπορεί η δυνητική έννοια εδώ ε, επιτρέπει και τη χρηματοδότηση της έρευνας βεβαίως το αποτέλεσμα της βασικής έρευνας και οι προοπτικές που θα δημιουργήσει δεν μπορούν να υπολογιστούν, δεν είναι προβλέψιμες. Ε, και σε μια εποχή όπου από οικονομική άποψη βρισκόμαστε σε άσκημη κατάσταση αυτό δεν είναι καλό και δεν μπορούμε να βασιστούμε στη βασική έρευνα με αυτή την έννοια. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Θα πρέπει να δούμε ολόκληρη την αλυσίδα από τη βασική έρευνα μέχρι την πραγματική εφαρμογή. Καλύτερες συνθήκες για εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, για ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων κτλ. Και αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να προχωρήσουμε. Η ολόκληρη αλυσίδα που την βασική έρευνα, με τα νέα προϊόντα που μπαίνουν στην αγορά πρέπει να μελετηθεί. Βεβαίω υπάρχει ένα κενό μεταξύ των πιλωτικών προγραμμάτων και των πρωτότυπων ε, ή μικρών, ε, αν θέλετε, πρώτων παραγωγών. Ωραία, υπάρχει αυτό το κενό ε, και πολλοί φωνάζουν ότι θα πρέπει να καλυφθεί, να γεφυρωθεί αυτό το κενό. Αυτό είναι η πρόκληση της νέας δεκαετίας, της επόμενης δεκαετίας. Μας λένε και στην Αυσία και στις Ηνωμένες Πολίτες και παντού. Αν όμως κοιτάξει κανείς αυτή την αλυσίδα που ανέφερα πριν, θα πρέπει να, θα συνειδητοποιήσουμε δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ βασικής έρευνας, εφαρμοσμένης έρευνας κτλ. κτλ. Τα πράγματα μπορούν να επηρεαστούν σε κάθε σημείο. Δεν είναι ε, νομοτελειακή η εξέλιξη της αλυσίδας αν θέλετε. Ανα πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί πρόσθετη προστιθέμενη αξία, να δημιουργηθεί μια καινοτομία, να και όχι μόνο ε, και νέες τεχνολογίες, όχι μόνο καινοτόμες, αλλά και τεχνολογίες που μπορούν να α, βελτιώσουν, που δεν είναι την κατάσταση και να οδηγήσουν σε νέους κλάδους, νέες αγορές. Θα δώσω ένα παράδειγμα αυτών των λεγόμενων transformative technologies. Ε, θα δώσω ένα παράδειγμα για τα, την μαγνητική τομογραφία στην, στα νοσοκομεία της Ευρώπης. Εκεί έγιναν αλλαγές τα τελευταία χρόνια που πραγματικά ε, οδήγησαν σε μια καινούρια κατάσταση που δεν μπορούσαμε να τη πριν από χρόνια. Ε. Ε, βεβαίως η εξέλιξη κάποιου αποτελέσματος βασικής έρευνας δεν μπορεί να μας οδηγήσει απαραίτητα ή δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν θα μας οδηγήσει στην α, β, γ τεχνολογία γι' αυτό η Ευρώπη θα πρέπει να χρηματοδοτήσει και να επενδύσει στις αναδυόμενες τεχνολογίες όποιες και να είναι αυτές δεν λέω ότι υπάρχουν βεβαιότητες εδώ είναι τελείως ε, αβέβαια τα πράγματα γι' αυτό μοιραία χρειάζεται μια ελαστική ανταπόκριση σε αυτά που συμβαίνουν και ταχύ ανταπόκριση όμως τι θέλω να πω με την περιγραφή αυτών των σενάριων. Ότι η Ευρώπη δεν είναι ένα απλό επίπεδο περιορισμένο πεδίο για τους Ευρωπαίους. Λέμε ότι βεβαίως δεν θέλουμε να υπάρχει προστατευτισμός, άρα δεν είμαστε κλειστοί, είμαστε ανοιχτοί. Αυτό δεν αρκεί όμως και πρέπει να γίνονται προσπάθειες για να πάμε πιο γρήγορα κτλ. Ναι βεβαίως, και κάποιες τέτοιες μεταβλητές έχουν ήδη προδιοριστεί, ανοιχτές αγορές, ανοιχτή προσέγγιση κτλ. Αλλά υπάρχουν και άλλες ε, ευελιξίες που πρέπει να έχει το σύστημα και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι να καθίσουμε να ξανασκεφθούμε από την αρχή τις επενδύσεις ε, και πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τα ρίσκα από τις επενδύσεις Εδώ μπαίνει το θέμα της Ευρω... του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεστιχνίας. Η Ευρωπαϊκή Πατέντα είναι απαραίτητη εδώ για αν θέλουμε να προχωρήσουμε τέλος ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι το εξή. Η κινητικότητα, η κινητικότητα των πολιτών, των ερευνητών κτλ. Βεβαίως ε, μπορούμε να οδηγηθούμε εδώ σε ένα, τη μια ενδοκινοτική τρόπον την ενδοευρωπαϊκή φυγή εγκεφάλων όπου θα έχουμε μια κίνηση της έρευνας προς την ανεπτυγμένη αν θέλετε ερευνητικά Δυτική Ευρώπη αυτό ε, θα πρέπει να το προσέξουμε και ε, παρόλα που στην Δυτική Ευρώπη υπάρχουν πολύ σημαντικές οργανώσεις ε, και δημόσιες όχι ιδιωτικέ, παρόλο υπάρχουν και ιδιωτικέ. Ε, στην Ολλανδία, παραδείγματο χάρη, είναι το Fraunhofer Institute που δουλεύω εγώ, είναι μια άλλη περίπτωση. Υπάρχουν πάντω αυτέ οι οργανώσει στην Ευρώπη, οι οποίε είναι ουσιαστικά το interface μεταξύ των μεν και των δε και γεωγραφικά και μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και παλιάς και νέας τεχνολογίας κτλ. Άρα θα πρέπει να προωθηθούν οι οργανώσεις αυτές. Ε, ε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε για να σας δώσω ένα παράδειγμα να φτιάξουμε ένα μικρό πρόγραμμα για πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτή είναι η απάντηση για το που θα βάζαμε το ένα δις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα οδηγούσαν σε σημαντικά αποτελέσματα Ευχαριστώ Πάτρικ Χωσέ Ευχαριστώ πολύ είχα προετοιμάσει το έγγραφό μου στα αγγλικά αλλά βέβαια ομιλείται η Πορτογαλική στο κοινοβούλιο αυτό και αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει την ευρωπαϊκή διαφορετικότητα. Αν έπρεπε να δώσω ένα τίτλο στην παρουσίασή μου, δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια, αλλά θα διάλεγα το εξής. Θα ομιλούσα για έξυπνη ανάπτυξη, μεν, αλλά μια έξυπνη ανάπτυξη ίσως και χωρίς ανάπτυξη. Τώρα αυτό ε, σαν φράση δεν λέει τίποτα, είναι κάτι το εντελώς αντιφατικό σαν διατύπωση. παρόλα αυτά έχει κάποιο νόημα. Γιατί έχει κάποιο νόημα. Θα ήθελα να μου δώσετε τη δυνατότητα να εξηγήσω το ότι σήμερα ζούμε σε μία κατάσταση όπου η ανάπτυξη φυσικά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο Και γι' αυτό αυτό το οποίο στην πρώτη φάση θα με απασχολήσει είναι η σχέση καινοτομίας και ανάπτυξης από την άλλη. Και σε ποιο βαθμό μια τέτοια σχέση μπορεί να είναι η ίδια σε διαφορετικά οικονομικά πλαίσια. Μπορούμε να πούμε ότι η καινοτομία είναι μια ισχυροτάτη μορφή ενέργειας που οδηγεί στην ανάπτυξη. Και το βασικό θα έλεγα αποτέλεσμα της καινοτομίας είναι η παραγωγή αποτελεσμάτων μεγάλου βάρους και μεγάλης εμβέλειας που επηρεάζουν το σύνολο της οικονομίας. Όταν μιλάμε λοιπόν για την καινοτομία, το θέμα δεν είναι να δούμε αν θα συνοδεύεται από την οικονομική ανάπτυξη και στην περίπτωσή μας τον τελευταίο καιρό από μια πολύ χαμηλή ανάπτυξη αλλά το αν η καινοτομία αυτή καλείται να παίξει ένα ρόλο που να γεννήσει στο μέλλον ανάπτυξη. Βλέπουμε ότι επηρεάζει η καινοτομία την ανάπτυξη, αλλά μέχρι τώρα την επηρεάζει σε τοπικό επίπεδο και επιμέρους μόνο η καινοτομία δεν λειτουργεί συνολικά, δεν εκμεταλλεύεται το μεγάλο της βάρος, δεν ξεπερνάει τον τοπικό χαρακτήρα και δεν διαφοροποιεί την κατάσταση και τις ασυμμετρίες παρά μόνο τοπικά και επηρεάζει έτσι την οικονομική δομή τοπικά και όχι σε εθνικό ή υπερεθνικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που ήθελα να κάνω, είναι ένα ερώτημα ουσιαστικά για το εάν το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο αναφερόμεθα είναι αποφασιστικό και μας βοηθά να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για τις σχέσεις ανάμεσα σε καινοτομία και ανάπτυξη. Η δεύτερη παρατήρηση ερώτηση. Θα πρέπει να δούμε αυτή η Ευρώπη, η ανεμική σε επίπεδο ανάπτυξης, τι αντιπροσωπεύει ε, πλέον σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια διαπιστωμένη πλέον ανεμία θα έλεγα. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρώπης σήμερα είναι η απασχόληση. Η δημιουργία δηλαδή των απαιτουμένων ε, συνθήκων οι οποίες θα βοηθήσουν στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και μείωση της ανεργίας. Σαν οικονομολόγος νομίζω ότι δεν υπάρχουν trade-off ανάμεσα στις επιχειρήσεις και την καινοτομία. Νομίζω επίσης ότι όταν και οι δύο αυτές παράμετροι και η καινοτομία και η απασχόληση εξαρτώνται από ένα παρόμοιο πλαίσιο, από ένα παρόμοιο περιβάλλον, από το ότι σαν παράδειγμα η οικονομία θα πρέπει να μπορέσει να κινητοποιήσει πλήρως το αναπτυξιακό της δυναμικό. Αυτό θα ήταν ο στόχος και αυτό δεν συμβαίνει στην Ευρώπη του σήμερα και γι' αυτό χαρακτηρίζουμε την Ευρώπη του σήμερα οικονομικά και αναπτυξιακά ανεμική. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας το σενάριο της αδύνατης Ευρώπης, της αδύνατης με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπάρξει η Ευρώπη όπως τη θέλουμε. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με την ανάγκη μιας ρήξης, μιας ρήξης ανάμεσα στις κεντρικές οικονομικές δυνάμεις στην παγκόσμια σκηνή και την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι αλήθεια ότι το μέγεθος ενός προϋπολογισμού δεν είναι πάντα κάτι το καθοριστικό. Αλλά είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που αντιπροσωπεύει το ένα του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ θα ήταν κάτι το επαρκές. Τέταρτη παρατήρηση να κάνω αναφορά σε, μια, σε έναν όρο που έχει εξαφανιστεί από το ευρωπαϊκό λεξιλόγιο τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια. Είναι ο όρος συνοχή. Όταν αναφέρομαι στη συνοχή, αναφέρομαι και στην εδαφική συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην κοινωνική συνοχή. Ένα από τα προβλήματα και ένας από τους στόχους του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι η εκ νέου εφεύρεση θα έλεγα αυτής της συνοχής μέσω επενδύσεων στις υποδομές και μέσω επενδύσεων στην καινοτομία, καθοριστική τομής και οι για την ευρωπαϊκή οικονομία. Εδώ θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση. Ίσως ζούμε μια περίοδο όπου οι υπερβολικές εξουσίες που δόθηκαν στις αγορές οδήγησαν στον θάνατο κάποιων δυναμικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς όπως δυστυχώς και στον τεχνολογικό και τον καινοτομικό γενικότερα τομέα. Η καινοτομία είναι ένας όρος λοιπόν που μας επιτρέψει να αναστήσουμε μια νέα απαραίτητη διάσταση για την οικονομία και με μια κοινωνική φυσικά σημαντική πλευρά. Το θέμα είναι βέβαια είναι ότι δεν θα ξέρουμε τι έχουμε ανάγκη σε τρία χρόνια. Μπορούμε ίσως σε τρία χρόνια να μιλάμε για την ευρωπαϊκή απεικοδόμηση. Και σε αυτή την περίπτωση ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να το αποφύγουμε. Μπορούμε να ζητήσουμε την ανικοδόμηση της Ευρώπης με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες. Ή χρειάζεται ο προϋπολογισμός και νέα στοιχεία, κάτι το οποίο μας οδηγεί στην έξυπνη μορφή ανάπτυξης που συζητάμε σήμερα. Και κλείνοντας να μου επιτρέψετε να σχολιάσω και την ερώτηση του ενός δις ευρώ. Την πρόταση που θα κάνω την έχουν κάνει πολλοί. Τα μισά λεφτά θα τα δώσω στο πανεπιστήμια και τα άλλα μισά λεφτά θα τα δώσω στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις οι οποίες θα εμπλακούν στην οδό της καινοτομίας και στην δημιουργία υψηλού επίπεδου θέσεων απασχόλησης. Και έτσι και τα πανεπιστήμια θα μπορέσουν και αυτά να δημιουργήσουν ε, προστιθέμενη αξία και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τότε μόνο θα μπορέσουμε να αναδείξουμε και την πραγματική διάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τύπο μαθηματικό που να καλύψει τις ανάγκες της οικονομίας αλλά και του κοινωνικού κεφαλαίου. Ευχαριστώ καθηγητά Ράις. Το λόγο έχει η κυρία Λέσλι Βίλσον από την Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντρέα, ευχαριστώ. Είμαι εκπρόσωπος μιας οργάνωσης που συνενώνει αρκετά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι τα πανεπιστήμια καλωσορίζουν τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και γιατί είναι σε καλή θέση ώστε να διαπιστώσουν ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, ε, των παγκόσμιων εξελίξεων. Θα δείτε τις κατατάξεις και τις αξιολογήσεις και θα δείτε πόσο συζητείται η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ε, και η προοδευτική φθήνουσα τάση και υπάρχουν και κάποια πανεπιστήμια από την Ασία τα οποία ανεβαίνουν. Και όλα αυτά συζητούνται στο πλαίσιο τη ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Ε, σε αυτό το πλαίσιο, η χρηματοδότηση της έρευνας, της καινοτομίας αλλά και της εκπαίδευση ε, της ε, διαβίου μάθησης, της κατάρτισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κινητήριος μοχλός σήμερα για τον εξυγχρονισμό ε, του όλου πανεπιστημιακού συστήματος από βορρά σε νότο και από ανατολή στη δύση, διότι παρέχει εργαλεία που θα ενισχύσουν τη διαδικτύωση, την ερευνητική συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων αλλά και μεταξύ πανεπιστημίων και εταίρων τους από τη βιομηχανία, τους δήμους, τις κοινότητες και αλλού ανά την Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο ώστε να βελτιώσουν και την ανταγωνιστικότητά τους δεύτερον παρέχει μηχανισμούς κινητικότητας ε, για τους νεαρούς Ευρωπαίους, αναφέρθηκαν κάποιοι από αυτούς, και στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών του σπουδών και πιο πριν. Και ενισχύει επίση και την ανταλλαγή ερευνητών ε, και σε επίπεδο διδακτορικού και μετά. Επίση παρέχει κατά τρίτον δυνατότητε για τη βελτίωση τη ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών στην Ευρώπη. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, αν λάβει κανεί υπόψη την ανάγκη βελτίωση τη απασχολησιμότητα ε, των αποφύτων, βελτίωση των δεξιοτήτων, ε, ό,τι μαθαίνουν δηλαδή όσου σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο. Και βέβαια έχουμε το το στόχο του 40% στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 και νομίζω ότι μαζί με την έρευνα και την καινοτομία η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η διαβημάθηση είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες. Δεύτερο σημείο, η έρευνα και η καινοτομία, η δημόσια χρηματοδότηση αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ίσως να είναι ούτε καν το 7% της χρηματοδότησης, πιστεύω ότι έχει σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, διότι κατά βάση παρέχει ε, ελεύθερη πρόσβαση ε, σε χρήματα ε, για τα πανεπιστήμια. Και σημαντικό ποσοστό των εθνικών κονδυλίων για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι για τις υποδομές στα κτίρια τους μισθούς. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί την εισαγωγή πολύ σημαντικών προγραμμάτων και βοηθά τα πανεπιστήμια να βελτιώσουν τα ισχυρά του σημεία και να προσφέρουν νέες δυνατότητες, νέες ευκαιρίες. Αυτό το παραβλέπουμε, γίνεται σήμερα στην Ευρώπη και με την ανταλλαγή ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις επιχειρήσεις μεταξύ άλλων και άλλους εταίρους. Τώρα, υπάρχουν κάποια εργαλεία που έχουν καθιερωθεί. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και να προτείνω βέβαια κάποια πρόσθετα εργαλεία. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο που αναφέρατε και το οποίο πραγματικά έχει κάνει τη διαφορά. Επίσης έχουμε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την πρόθεση της ανταγωνιστικότητας στη βασική έρευνα. Δεύτερον, διάφορα προγράμματα συνεργασίας που επίσης είναι σημαντικά για να υπάρχει συμμετοχή των πανεπιστημίων στο πρόγραμμα πλαίσιο συνένωση ερευνητικών ε, ομάδων, εξωτερικούς εταίρου σε σημαντικούς ερευνητικούς τομείς που θα ανταποκριθούν όλο και περισσότερο στις βασικές προκλήσεις για τον τομέα της ενέργειας, για παράδειγμα, όπου γίνεται σημαντική προσπάθεια στο επίπεδο των πανεπιστημίων. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την κοινή ανάπτυξη και εκπόνηση προγραμμάτων ε, και ε, προγραμμάτων σπουδών. Η δράση Marie Curie επίσης ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό, έχει διάφορα στοιχεία και μέσα σε αυτά είναι και η ενίσχυση της καινοτομία. Το πλαίσιο των δράσεων των μέσων που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα και για το μέλλον και για να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τη μετοχή των πανεπιστημίων στην ευφύ ανάπτυξη, νομίζω ότι καλό θα ήταν ίσως να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε συνεργασίες μεταξύ παραδείγματος χάρη διαφορετικών στοιχείων και σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, την ενία αγορά. Έχουμε την ε, πρόταση για την αναθεώρηση οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία, νομίζω, για την Ευρώπη για να κάνει πραγματικά τη διαφορά σε σχέση με τη μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση μάλλον αυτή τη οδηγία και τη διασύνδεσή τη με την κινητικότητα και του στόχου τη κινητικότητα. Παραδείγματο χάρη, να διασυνδεθεί αυτό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και την υλοποίησή του, τη σημασία που έχει να προωθήσουμε περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα την κατάρτιση την ατυπική μάθηση, ε, την εκπαίδευση, την κατάρτιση σε σχέση με την ανάπτυξη του, διαβατηρίου, ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου προσόντων. Ο ρόλος των πανεπιστημίων ε, είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε ε, και την αναπτυξιακή ατζέντα που και εκεί μπορεί στην ανάπτυξη δηλαδή να κάνει κάποιο το πανεπιστήμιο. Επίσης, πέμπτον, όλα τα προγράμματα χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια ε, έχουν ένα σημαντικό στοιχείο, την απλούστευση για να μειωθεί το άχθος στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στα οποία μπορώ να επανέλθω. Και τέλος, για να απαντήσω και εγώ στο ερώτημα του ενός δις, έτσι δίνοντας και μια ευχάριστη νότα στο τέλος της πρώτης συζήτησης, είναι πολύ απλή η πρόταση του Αντρέ Σαπίρ ε, και εμείς το ίδιο κάνουμε. Παραλλήλου έχουμε λοιπόν ε, μια πρόταση επιτάπητος, την έχουμε υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Ρημπτικό Συμβούλιο ε, για ανταγωνισμό των μεταπτυχιακών, των σχολείων που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα, διεκτορικό συγκεκριμένα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Θα ήταν σημαντικό να υπάρχουν υποτροφίες μέσω αυτού του Συμβουλίου για υπηκός τρίτων χωρών, ώστε η Ευρώπη πραγματικά να μπορεί να εκπονήσει σημαντικά διεθνή προγράμματα. Έχουμε τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, να βοηθήσουμε επίσης να υπάρχει και μεγαλύτερη ερευνητική δυνατότητα ε, και ανταγωνιστικότητα σε αυτή την παγκόσμια αγορά ταλέντων. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Λέσλι. Κλείνει εδώ, νομίζω, ο κύκλος ο πρώτος κύκλος παρεμβάσεων, ακούσαν πολλές ιδέες, πολλές προτάσεις. Τώρα λοιπόν θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο σε εσά, στους ευρωβουλευτές. Για να δούμε ποιος θέλει το λόγο. Εγώ, εγώ, Σαλβαντόρ, Ταρίκα, Γκάρια Ζαμπάλ, Derek Βόν... Έχω πολύ μεγάλο κατάλογο μιλητών. Ε, Derek Warren, Josie Lewis. Äh, ε, ε, Ο εισηγητής μας όμως πρέπει να αρχίσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως και ο κύριος ε, Ρέις, θα εκμεταλλευτώ και εγώ τη δυνατότητα της ταυτόχρονης διερμηνίας και θα μιλήσω και εγώ τη μητρική μου γλώσσα. Παρέμβαση του κυρίου Σαπίρ, θέτει κάποια σημαντικά ζητήματα. Νομίζω βέβαια ότι μία από τις ε, φράσεις που θα μπορούσε να ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο, όπως και ο κύριος Ρέης, είναι ότι εδώ ε, αποσυναρμολογούμε ή επαναφευρίσκουμε ή επανανακαλύπτουμε την Ευρώπη. Είναι το ζήτημα που συζητούμε και σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Φοβάμαι ότι μήπως αποσυναρμολογούμε, διασπούμε τελικά την Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για τη στρατηγική 2020 τόσο στον ιδιωτικό τομέα και πιστεύω και εγώ και στον δημόσιο τομέα υπάρχουν επίσης ε, κάποιες αμφιβολίες. Η στρατηγική 2020 προϋποθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσεις ε, που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιήσει κανείς, που είναι δεσμευτικές. Αλλά νομίζω ότι είναι προφανές ότι αυτό που έχει ανάγκη ο ιδιωτικός τομέας είναι πίστη. Επομένως, από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που πρέπει να δώσουμε ε, στον ιδιωτικό τομέα είναι η πίστη, η χρηματοοικονομική πίστη και όσο τον πιο γρήγορα. Τώρα, ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σαπίρ το εξή. Τι είναι πραγματικά η καινοτομία, γιατί μιλάμε για καινοτομία και εγώ νομίζω ότι τελικά η καινοτομία είναι ένα εργαλείο και ο τελικός ε, σκοπός είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας ε, των διαδικασιών παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι ο κοινοτικό προπολογισμό θα έπρεπε να χρησιμεύσει για να χρηματοδοτεί τα εργαλεία, τα μέσα και όχι τους στόχους. Εξού λοιπόν ε, θεωρώ ότι η καινοτομία θα έπρεπε να είναι ένας στόχος προτεραιότητας που θα χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προπολογισμό. Ο προβολισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλήσατε για τη βέλτιστη διάσταση, ποιο είναι το ιδανικό μέγεθο του κοινωτικού προπολογισμού. Θεωρείτε ότι το 1% πιστώσεων πληρωμών είναι το ιδανικό μέγεθος για τον κοινωτικό προπολογισμό και είναι εφικτό να γίνει κάτι σε κοινωτικό επίπεδο με αυτό το ποσό. Επίσης, ε, μιλάτε για την ευφυΐα των κρατών μελών. Η ευφυΐα των κρατών μελών, από ό,τι φαίνεται, ε, την εφαρμόζουν την ευφυΐα του στη μείωση του κοινωτικού προπολογισμού. Δεν ξέρω αν σε αυτό είναι πολύ ευφυής ε, και αν αυτό συνάδει με το ευρωπαϊκό μέλλον. Και δεν ξέρω αν ένας μικρότερος προπολογισμό σε μέγεθο θα ήταν και βιώσιμος. Και η πιο έτσι διαφιλονικούμενη δήλωση που κάνατε και που φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί είναι το θέμα της αριστείας. Η αριστεία στην καινοτομία, στην ανάπτυξη. Τελικά η καινοτομία είναι ένα μέσος ε, διάθεσης, κατανομής γλίσχρων οικονομικών πόρων. Είναι ένα δημοσιονομικό εργαλείο δηλαδή. Στην πράξη όμως, πρώτον, μπορεί να υπάρχει καινοτόμος προϋπολογισμός, προϋπολογισμός καινοτομίας που να συνενώνει, να περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό, το μεγαλύτερο μέρος των εθνικών προϋπολογισμών για την καινοτομία. Εσείς λέτε ότι η καινοτομία φαίνεται από την αριστεία και την ανταγωνιστικότητα. Αυτό όμως ε, έχει αντικρουστεί. Υπάρχει και μία έκθεση την οποία αναθέσαμε εμείς στην Επιτροπή μας και που δείχνει ότι σήμερα σε ό,τι αφορά την καινοτομία το μέρος της ε, ανταγωνιστικότητας χρηματοδοτείται από την κατηγορία 1β κατά κύριο λόγο στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, την κατηγορία της συνοχής δηλαδή. Η εφαρμογή λοιπόν της αριστείας υπό την αυστηρή του όρου θα μας οδηγούσε ίσως στο στην εξή κατάσταση η συνοχή να χρηματοδοτεί σήμερα την πολιτική καινοτομία. Και αυτό, όπω είναι προφανέ, πρώτον δημιουργεί προβλήματα και αντιπαθέ. Δεύτερον, αφαιρεί ε, την αρχή τη επικουρικότητα. Και τρίτον, δεν θα υπήρχε αναδιανεμητικό προπολογισμό. Τι αναλλακτικέ λύσει έχετε να προτείνετε εσεί. Και τέλο, ένα ερώτημα προ την κυρία Νίλσεν. Μιλάμε για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Νομίζω ότι το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο αρχίζει λίγο πολύ πριν να έχουν σχεδιαστεί οι προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές. Εσείς ε, πώς θεωρείτε ε, ότι αυτό το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριλάβει στρατηγική 2020. Μέσω της 2020 όπως προτείνει και η Επιτροπή 2020 ή πρέπει να υπάρχουν και άλλοι στόχοι. Ähm, der Berichterstatter hat jetzt etwas länger reden dürfen. Ich muss... Ο εισηγητής μίλησε λίγο παραπάνω. Του δίνουμε αυτό το δικαίωμα. Αλλά για τους επόμενους ομιλητές θα είμαι πιο αυστηρή. Eh, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να εκφραστώ στην πορτογαλική γλώσσα. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω και να σας συγχαρώ για την ποιότητα των παρεμβάσεων σας, λέει ο κ. Φερνάνδης. Να μιλήσω τώρα για τα πρότυπα, τα οποία εμείς τα επιθυμούσαμε έτσι ώστε να οδηγηθούμε στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο για ε, την ε, ε, ανάπτυξη και την έρευνα. Ένα το οποίο θα καθορίζει εκ των άνω προς τα κάτω τα διαθέσιμα ποσά ή μήπω θέλουμε ένα πρότυπο εκ των κάτω προς τα πάνω το οποίο θα καθορίζει γενικούς στόχους και η προσθεσή τους θα συναποτελεί το τελικό ποσό. Η έξυπνη ανάπτυξη, και αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, είναι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να δώσουμε μια απάντηση στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Για να παρουσιάσω περιληπτικά την στρατηγική 2020, να πω ότι στοχεύει στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να προέλθει από μια έξυπνη ανάπτυξη, ίσως περιορισμένη αριθμητικά, η οποία ονομάζεται αηφόρος ουσιαστικά ανάπτυξη. Και εδώ σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς αυτό που ονομάζουμε έξυπνες μορφές ανάπτυξης. Αν κατάλαβα καλά θα μπορούσαμε να έχουμε στη διάθεσή μας ένα ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο οποίος να είναι αποσυνδεδεμένος από τα εθνικά δημοσιονομικά σχέδια. Δεν ξέρω, ίσως παρεμεινεύω τον κύριο Σαπίρα, αλλά ίσως ταυτόχρονα δεν είναι απαραίτητο αυτός ο σύνδεσμος. Είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι κάτι το υποχρεωτικό. Το διαπιστώνουμε και στις πράξεις μας, στις δράσεις μας, συγγνώμη, στους στόχους τους οποίους καθορίζουμε και διαπιστώνουμε ότι πράγματι πρέπει να υπάρξει ο ανταγωνισμός αυτός και διαρωτώ με ποιες είναι οι προτάσεις που κάνετε έτσι ώστε οι συντονισμοί αυτοί ενώ οι μορφές συντονισμού ανάμεσα στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στους εθνικούς προϋπολογισμούς σε όλους τους τομείς της στρατηγικής 2020. Ιδιαίτερα όμως στον τομέα όπου έχουμε τα 500 εκατομμύρια και αυτήν την τεράστια αγορά ικανότητας και ταλέντου. Είναι, είναι κρίμα ορισμένα είναι τραγωδία ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν και όπου έχουμε απλώς καταναλωθέν χρήμα και όχι επενδεδημένο χρήμα από τον προϋπολογισμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Υπάρχουν πιέσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ορισμένα πράγματα και να λογοδοτήσουμε. Ρωτώ λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να, ε, για να ξοδε, οι δαπάντες, ώστε οι μας να πηγαίνουν σε πραγματικά καλές επενδύσεις, νόμιμες και καλές επενδύσεις και εγώ νομίζω ότι η ευρωπαϊκή κρίση είναι μια ευκαιρία για να αλλάξουμε και ορισμένα πράγματα γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ορισμένα ε, βλέπουμε ότι οι κακοί μαθητές παίρνουν πολλά χρήματα. Δηλαδή η Νότια Ιταλία η οποία έχει σωρό προβλήματα ε, βλέπουμε να χρηματοδοτείται συνεχώς. Πώς μπορούμε λοιπόν να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση η οποία δεν εξυπηρετεί κανένα νομίζουμε. Ε, uh, <coughs> Ευχαριστώ. Μία ερώτηση για όλους τους ομιλητές. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας, μιλήσατε για μια σκεπτικιστική ε, αντίληψη. Είπατε κύριε Σαπρί στην αρχή ότι δεν ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του κόσμου η στρατηγική τη Λισαβόνα η εφαρμογή τη, αλλά φαίνεται για την άλλη στρατηγική, τη στρατηγική 2020, να είστε πολύ πιο αισιόδοξοι. Ποια είναι η διαφορά, τι διαφέρει αυτή η στρατηγική από την προηγούμενη τη Λισαβόνα, τι συνέβη δηλαδή, Είναι οι στόχοι ή το πρόβλημα, οι μέθοδοι, τα μέσα, οι τομεί, που θα επενδυθούν τα χρήματα. Εμείς είμαστε πολιτικώς αισιόδοξοι, εσείς είστε όμως οι εμπειρογνώμονες. Γιατί είστε εσείς τόσο αισιόδοξοι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ Λισαβόνας και 2020. Βέβαια γίνεται μια εκ των προτέρων αξιολόγηση, αυτή που σας ζητώ τώρα να κάνετε. Είναι μια εξάντε αξιολόγηση. Επίσης, ο πρόεδρος ε, Σαπίρ ε, που γνωρίζω το έργο σας είπατε κάτι, είπε κάτι πολύ ε, ξυπνό για τα κριτήρια της αριστείας, γιατί είπατε ότι τα άλλα έχουν τους δικούς τους πόρους. Εμείς είμαστε η προοπτική για τους δημοσιονομικές προοπτικές, όχι για ό,τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή και σε εθνικό επίπεδο, αλλά εδώ γίνεται μια πολύ σημαντική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι καλύτερο στη στρατηγική 2020, να υπάρχουν νέε προτεραιότητε όπως αυτό που είπατε, ευφυείς, βιώσιμη για όλους. Ή όλες οι πολιτικές λαμβάνουν υπόψη σε, τις προτεραιότητες σε κάθε πολιτική καινοτομία, ευφυή, βιώσιμη κτλ. Συνοχή, το ίδιο, ευφυείς, βιώσιμη για όλους. Ή μήπω είναι καλύτερο, που είναι και η σημερινή τάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισήμως στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού, να γίνει κάτι τομεακό. Δηλαδή βάζουμε κάποιες ε, στο ευφυεί πολιτικές, κάποιες άλλε πολιτικέ τι βάζουμε στο για όλους και κάποιες άλλες βάζουμε στο βιώσιμη. Τι είναι καλύτερο να κάνουμε όμω. Ε, και ε, γι' αυτό λοιπόν θέλω την άποψή σα και για τη διαφορά Λισαβόνα 2020 και για το αν θα θέλουμε να το τομεοποιήσει οριζόντια προέλευση. Ευχαριστώ. Η επόμενη συνάδελφος, Καρδιά Θάμπαλ. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Ρέντα, όταν έκανε την εισαγωγή του, είπε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά ε, την επένδυση πόρων για την καινοτομία και την έρευνα από το δημόσιο κορβανά δεν τα πάμε και τόσο άσχημα, αλλά σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό σκέλος ε, εκεί δεν τα πάμε καλά σε σχέση με μεγάλες δυνάμεις όπως είναι παραδείγματος χάρη όπου η επιχειρηματική ε, τάξη αυτή ουσιαστικά είναι στην πρώτη γραμμή. Γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά και πώς θα μπορούσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον δικό μας τον προϋπολογισμό έτσι ταπεινά να αλλάξουμε την ισορροπία αυτή. Δεύτερο ερώτημα κάτι σε σχέση με αυτό που είπε και προλαλή σα, Ποια είναι η διαφορά της Αττικής 2020, γιατί μπορούμε τώρα να είμαστε αισιόδοξοι ή πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα σφάλματα του παρελθόντος, ε, γιατί όπως είπε ο κύριος Σαπέρ, φυσικά και δεν μπορούμε να χάσουμε άλλα 10 χρόνια, ε, ούτε και πριν βέβαια θα, μπορούσε, ήταν καλό να το είχαμε κάνει, αλλά είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε σήμερα. Επίσης, μιλήσατε για το μέγεθος των προπολογισμών και θα ήθελα οι εμπειρογνώμονες ε, να ε, τολμήσουν λίγο, να πάρουν ένα ρίσκο και να μας πούν ποιο είναι ε, για κατά αυτούς το βέλτιστο ποσοστό και σε ποια κεφάλαια θα έπρεπε να επενδύσουμε. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Επομένουν τρεις ακόμη συνάδελφοι που θα πάρουν το λόγο και μετά θα δοθούν οι απαντήσει από το πάνελ. πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. για το αν θα πρέπει να βασίζεται η οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καινοτομία και στη γνώση. Δεν ξέρω πού είναι εκεί η θέση ε, της επένδυσης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Απαιτείται να υπάρξει όμως και μια στενότερη σχέση ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο και τον ακαδημαϊκό κόσμο. Έχουμε κάποια θετικά παραδείγματα από την Ουαλία και σαν αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας κάποια νέα ε, πολύ ενδιαφέροντα προϊόντα κυκλοφορούν στις αγορές. Αλλά αυτό γίνεται με πολύ αργό τρόπο και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στον ακαδημαϊκό κόσμο και τις επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομία στο μέλλον. Η δεύτερη σχετικά με το fpa 8 όλοι μπαίνουμε αυτή τη στιγμή σε μια νέα α, περίοδο. In the future it works better for everyone. Τι θα γίνει με το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ja, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, dass mir die bisherigen Wortmeldungen θα ήθελα να πω ότι μέχρι τούδε παρεμβάσεις μου φάνηκαν υπερβολικά γενικές. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε με τις πολιτικές προτεραιότητες και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες, τις δυνατότητες του προπολογισμού. Αν κατάλαβα καλά, τι είπατε, είπατε ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Για το 2011, τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις, τι γίνεται η Ιρλανδία, πώς επηρεάζει το μέλλον, η ασπίδα προστασίας πώς επηρεάζει το μέλλον. Δεύτερο, μιλάμε για έρευνα. Έχει, υπάρχει δυναμικό και ικανότητες έρευνα στην Ευρώπη. Η στρατηγική του 2020 σε τελευταία ανάλυση δεν είναι οικονομικό ζήτημα. Είναι πολιτικό θέμα που Α, ουσιαστικά πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε πού χρειάζεται να μετατοπίσουμε κάποιες ικανότητες ερευνητικέ σε ποιους τομείς. Τρίτο θέμα, η Ευρώπη θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ να Ε, θα πρέπει να προσέξει τι θα κάνει στο μέλλον τι έχει κάνει μέχρι τώρα και τι θα κάνει στο μέλλον πρέπει να παραμείνει αξιόπιστη γιατί τόσοι πολλοί ερευνητές ε, λένε ότι είναι πολύ γραφειοκροτικά τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά και γι' αυτό δεν ε, οδηγούν σε αποτελέσματα εκείνο μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε καλά αποτελέσματα και όχι να έχουμε την έρευνα απέναντί μας ή φυγή εγκεφάλων Ευχαριστώ Δύο ερωτήσεις. λέει κυρία Τρούπελ, ακούσαμε στην αρχή της συζήτησης ότι ε, την περασμένη δεκαετία, τούτη τη δεκαετία, στόχος μας ήταν ο, ο ανταγωνισμός. Ε, δεν επιτύχαμε τους στόχους μας. Η δεκαετία αυτή όμως η επόμενη αναφέρεται στην έξυπνη φιλόσοφη ε, βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Ρωτώ, βιώσιμη ανάπτυξη είναι ευκαιρία για έξυπνη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Και να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ντρέσλερ. Είπατε ότι αυτό το περίφημο ένα δις θα το εμφαν, ε, επενδύατε στις πολύ μικρές επιχειρήσεις για έρευνα κτλ. Και ερώτηση... Και γιατί δεν το κάνετε, γιατί δεν μπορεί να το κάνει η Ευρώπη. Χρόνια ολόκληρα μιλούσαμε για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλούμε για την καινοτομία. Έχουμε το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας Πού, γιατί απέτυχε λοιπόν η Ευρώπη, τι θα έπρεπε να έχει κάνει καλύτερα για να επιτύχει. Czy są możliwe wspólne cele przy tak zróżnicowanej Unii Europejskiej po jej rozszerzeniu? E, Νομίζω ότι ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ποικιλότητα, ιδιαίτερα μετά τη διεύρυνση. Αυτό πρέπει να μην το αγνοούμε. Η στρατηγική στόχη της Ευρώπης του 2020 πρέπει να δούμε αν είναι σαφώς ευκρινής. Έτσι τότε θα μπορέσουμε να τους πετύχουμε στο μέλλον. Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για κοινού στόχους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπω θα πρέπει να μιλήσουμε για το συνδυασμό των εθνικών μόνο απλά στόχων. Τρίτον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε σε ποιο βαθμό οι κοινοτικοί στόχοι θα μας επιτρέψουν να ακολουθήσουμε μία πορεία η οποία να είναι σχετικά βέβαιη και ε, τουλάχιστον εν μέρη προδιαγεγραμμένη και να μην περιμένουμε τις κατευθυντήριες γραμμές να έρθουν σε κάποια φάση της πορείας αυτής. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο τίθεται άμεσα, είναι ο καθορισμός των μεγάλων στρατηγικών γραμμών σε σχέση με τη σημερινή συγκυρία, σε σχέση με τις σημερινές συνθήκες. Οι σημερινές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν την επιδίωξη μακροπρόθεσμων στόχων γιατί υπάρχουν άμεσα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την κάλυψη της συγκυρίας. Και τέλος, η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται στην ε, συνδυαστική της δυνατότητα, στην ενιαία αγορά, στις κοινέ δράσεις ή μήπως οφείλεται στο ότι έχουμε έναν κοινό προϋπολογισμό, μικρό μεν, αλλά κοινό πάντα. Τελευταία ερώτηση. Έχω την αίσθηση ότι την εποχή της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να λειτουργήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, σε επίπεδο κλίμακας. Το κάνουμε αυτό στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Ευχαριστώ. Και τώρα τελείω, τελευταία η Μαρία Καβάγιο. To draw the attention of the colleagues and the participants of this hearing of the... Ναι. πιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στο, στην έκθεση που μόλις, ε, ε, που εγκρίθηκε για την ε, απλοποίηση των ε, διατάξεων και των ε, κανόνων συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα. Ε, 70 περίπου συστάσεις γίνονται για την απλοποίηση ε, για ούτως ώστε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να συμμετέχουν. Ε, είναι επίγον κατά την άποψή μας να εφαρμοστούν όλα αυτά και όπως ελέγχθηκε στην αρχή το πιο σημαντικό για μας είναι η εφαρμογή σε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένων ωραίων ε, ιδεών και και αν η στρατηγική ε, αν ε, τελικά η εφαρμογή είναι καλή θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αντίστοιχα πράγματα και σε άλλους τομείς. Ευχαριστώ. Thank you for all these comments. Uh, I hope that we will find the... Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Μακάρι να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Πάντως ε, είναι πολύ καλό σημάδι ότι όλοι είχατε πολύ επικοδομητικά σχόλια και ερωτήσεις. Ε, το Κοινοβούλιο πολλές φορές ε, απαντάει ε, πριν τεθούν τα ερωτήματα, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε και εμεί κάτι να πούμε. Θα ξεκινήσω ανάποδα αυτή τη φορά, δηλαδή με την τελευταία ομιλήτρια πρώτη, τη Λέσλι Wilson, η οποία μπορεί να σχολιάσει κάποια από ε, τα ερωτήματα που την αφορούσαν ή που τέθησαν σε όλους τους ομιλητές του πάνελ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα επικεντρωθώ στο ζήτημα του προγράμματος πλαισίου κυρίως. Θα επαναλάβω αυτό που είπε ο τελευταίος ομιλητής. Σε αυτή τη συζήτηση για την απλούστευση των διαδικασιών συμμετέχουμε και εμείς. Είναι σημαντικό για τα πανεπιστήμια αυτό. Απαντώντας λοιπόν στο ερώτημα γιατί δεν θέλουν πάντοτε τα πανεπιστήμια ή γιατί δεν μπορούν συχνά να λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα πλαίσιο, νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό γιατί είναι πολύ αναλυτικά τα ζητήματα. Πολλές φορές ε, ίσως να μην τόσο ελκυστικό θέμα, αλλά κάνει και τη διαφορά τελικά σε ό,τι αφορά τη διάθεση και τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων των προγραμμάτων πλαίσιο. Τι περιμένουμε τώρα ε, σε σχέση με το μέλλον, τι θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα δεδομένων των συνθήκων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας βαθμός συνέχειας ε, των εργαλείων από το ένα πρόγραμμα πλαίσιο στο άλλο. Νομίζω ότι εν γέννη, ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι σημαντικό να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα μέσα και προγράμματα αυτά τα οποία θα προκρίνουμε, παρότι μπορεί να είναι διαφορετική εστίασή τους θα πρέπει η επικάλυψη μεταξύ των διαφόρων εργαλείων να αποφεύγεται και πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχε πληθώρα αλληλοκαλυπτόμενων μέσων. Παραδείγματο χάρη, για εμά, είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα ε, πραγματικά είναι μια σαφή περίπτωση ενό ε, εργαλείου στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου που δίνει μεγάλη όθηση, μοναδική όθηση στα πανεπιστήμια. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Τεχνολογία από την άλλη, το οποίο όμω ακόμη δεν έχει αποδείξει ότι αποτελεί προστιθέμενη αξία. Ε, υπεράνω άλλων οργανώσεων όπως είναι οι Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές ε, Πρωτοβουλίες, οι κοινοπραξίες ε, και οι εταιρικέ σχέσεις στο πλαίσιο Marie Curie. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη και της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων. Και για να απαντήσω συντομία το θέμα των ιδιωτικών επενδύσεων, νομίζω ότι το ζήτημα είναι ότι χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις, βιώσιμες αηφόρε δημόσιε επενδύσει για την πρόθεση και των ιδιωτικών επενδύσεων. Και νομίζω ότι αυτό εξακολουθεί να είναι η βάση της ε, δυνατότητα έρευνα και καινοτομία των πανεπιστημίων και τη δυνατότητα συνεργασία του με εξωτερικού εταίρου. Εάν οι συνθήκε πλαισίου είναι υπερβολικά πολύπλοκε και γραφειοκρατικέ, που ίσω να γίνουν έτσι με τι κοινέ πρωτοβουλίε προγραμματισμού, θα πρέπει να βοηθήσουμε να είναι παραγωγικά τα πανεπιστήμια και άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί. Ευχαριστώ, καθηγητής Ρέις. Ε, Μια πρώτη παρατήρηση. Να υπογραμμίσω και αυτή την αναφορά η οποία έγινε στη διαδικασία απλοποίησης για την πρόσβαση σε ερευνητικά προγράμματα παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συνέλεξα πολλές πληροφορίες στις προσπάθειες που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις οποίες αναφέρθηκε η κυρία Καρβάλιο. Έχω την αίσθηση ότι η προσπάθεια που έγινε ήταν πολύ σημαντική. Το πρόβλημα της ποιότητας της έρευνας είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και πολλές φορές δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας, ακριβώς όμως λόγω κανόνων που καθιστούν την πρόσβαση στην έρευνα ιδιαίτερα δύσκολη. Αυτό είναι ο λόγος λοιπόν για τον οποίο υπάρχουν εξαιρετικές επιδόσεις οι οποίες παραμένουν ακόμα κρυφίες και προς ανακάλυψη, ενώ οι ικανότητες αυτές και οι γνώσεις αυτές θα μπορούσαν να έλθουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα εδώ πρόσβαση στην έρευνα, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε να βελτιώσουμε. Τώρα για αυτό θα βοηθήσει και στην γεφύρωση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας με τη στρατηγική 2020. Έχουμε μία έντονη τάση να διαπιστώνουμε στις δύο αυτές στρατηγικές τα ίδια προβλήματα. Ενώ πάρα πολύ συχνά δεν υπάρχουν ε, οι ίδιοι εταίροι Νομίζω ότι τα προβλήματα τα οποία επιβάλλονται λόγω του μεγέθους τους δείχνουν τα κενά τα οποία υπάρχουν και χαρακτηρίζουν την καθημερινή ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Οργάνωση. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει τα προσαρμοσμένα κατάλληλα επίπεδα συντονισμού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα σωστό συνδυασμό ανάμεσα στην οικονομική σφαίρα, την οικονομική ιδιωτική και την οικονομική δημόσια, την κοινωνία των πολιτών, τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτή τη στιγμή η απουσία ορισμένου ρόλου των συγκεκριμένων εταίρων ε, δημιουργεί συγχύσεις ε, και ιδιαίτερα οδηγεί στη σύγχυση των στόχων των δύο διαφορετικού τύπου, όπως είπαμε, στρατηγικών. Για την τελευταία ερώτηση θα συμφωνήσω λέγοντας ότι η αηφόρος ανάπτυξη είναι μια ευκαιρία για την δημιουργία μιας έξυπνης μορφής οικονομικής ανάπτυξης και αυτό για ένα απλό λόγο. Η λογική της οργάνωσης των οικονομιών της αηφορίας, των οικονομιών που σέβονται το περιβάλλον, των οικονομιών που σέβονται τις ικανότητες θα μπορέσουν νομίζω να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα οποία διαπιστώνουμε και τα προβλήματα που έχουμε στον τομέα και της καινοτομίας και της απασχόλησης. Υπάρχουν θέσεις απασχόλησης οι οποίες είναι ενδογενείς στην αηφορία και θα πρέπει να δημιουργηθούν και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης που εξαρτώνται ιδιαίτερα από την ίδια την καινοτομία. Και σχετικά με τα πρότυπα και τον συσχετισμό ανάμεσα στον κοινοτικό προϋπολογισμό και τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Εδώ δεν νομίζω παρά μόνο ε, μπορούμε να προτείνουμε την αναφορά ανάμεσα στη συμπληρωματικότητα των δύο προϋπολογισμών, των δύο τύπων προϋπολογισμών. Αυτή η συμπληρωματικότητα μας οδηγεί στην εφαρμογή της παλιάς καλής αρχής της επικουρικότητας. Ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος για την σωστή αξιοποίηση του ευρωπαϊκού επίπεδου eu encontro-me indiscutivelmente. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά. Εγώ βρίσκομαι από την πλευρά αυτών που πιστεύουν ότι το θέμα του προϋπολογισμού δεν είναι μόνο θέμα μεγέθους. Esta situação insustentável de uma Europa com ruptura. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μια Ευρώπη με διαρθρωτικές βαθιές ρογμές. Μια Ευρώπη η οποία να έχει ένα προϋπολογισμό που θα καλύψει τα κενά και τις ρογμές αυτές. Ευχαριστώ καθηγητά Ρέις. Ο κύριος Μπρέσλερ έχει το λόγο. Σας έθεσαν αρκετές ερωτήσεις κύριε Μπρέσλερ, βασικά μία ερώτηση αλλά μπορείτε να αντιδράσετε και στις άλλες. With the SBR business. There's, um, but this all fits into a whole picture that I have. Σε σχέση με την εικόνα. Obstacles are the... Τα εμπόδια είναι η απόδοση των επενδύσεων ε, για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου δεν είναι το ίδιο στην Ευρώπη σε σχέση με τη ΣΥΠΑ ή αλλού υπάρχει έλλειψη κοινών προτύπων. Εάν έχετε μια επιχειρηματική ιδέα, ένα ερευνητικό προϊόν ή αποτέλεσμα εφαρμοσμένη έρευνα και θέλετε να το διαθέσετε στην αγορά, να το φέρετε στην αγορά, αντιμετωπίζετε διαφορετικά πρότυπα, διαφορετικέ ρυθμίσει και κανονισμού σε καθένα κράτο ε, μέλο παρά το ότι υπάρχει αναρμόνιση. Πάντω ε, υπάρχουν αρκετά ακόμη που πρέπει να γίνουν για να υπάρχει συμβατότητα. Η άλλη ιδέα τώρα για το SPIR, ένα τέτοιο είδους ε, πρόγραμμα, η υποτροφία καινοτομία, αν θέλετε μπορούμε να το αποκαλέσουμε, αυτό είναι ό,τι πιο κοντά μπορώ να φανταστώ για να καλυφθεί αυτό το χάσμα καινοτομία. Η κοιλάδα θανάτου είναι η εξή. Πρέπει κανείς να ξεκινήσει παραγωγή μικρής κλίμακας και είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα γιατί αφήνει κανείς ε, τον ε, τομέα δημόσιας χρηματοδότησης και πηγαίνει στην ιδιωτική χρηματοδότηση και υπάρχει και μια γκρίζα ζώνη σε σχέση με τους ε, κανονισμούς με τις νομικές διατάξεις και τελικά καταλήγει κανείς με μια μεικτή χρηματοδότηση ενώ όμως χρειάζεται σαφής διαχωρισμός και ορισμοί γιατί αλλιώς μπορεί κανείς να κατηγορηθεί για κατάχρηση κεφαλαίων μεταφορά ή μια εγγραφή του στον προπολογισμό. Τώρα, σε αυτό το πολύπλοκο πλαίσιο πώς θα συνεργαστεί ε, ο ακαδημαϊκός κλάδος με τη βιομηχανία. Υπάρχει το IT, υπάρχει η τεχνολογία, αλλά όπως είπε και η Λέσλι, είναι λίγο πρόωρο να κάνει κανείς ε, μία δήλωση. Εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά είναι η επανεφεύρεση του τροχού. Αλλά ε, σίγουρα υπάρχουν οργανώσεις εφαρμοσμένης ε, έρευνας, υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο, πρόκειται για οργανώσεις εθνικές, οι οποίες ασχολούνται ακριβώς με το πρόβλημα αυτό. Πώς δηλαδή κανείς να ξεκινήσει μια μικρή επιχείρηση, πώς τα ερευνητικά αποτελέσματα των εφαρμοσμένων προγραμμάτων να τα εκμεταλλευτεί στις εταιρείες. και είναι πολύ πεπειραμένοι οι οργανισμοί αυτοί και σε ό,τι αφορά ε, τον εθνικό προπολογισμό και ίσως θα έπρεπε να δούμε τι κάνουν, τι κάνουν αυτές οι εθνικές οργανώσεις. Έπειτα, σε ό,τι αφορά το EIT, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας δηλαδή, ο στόχος του ίσως κάποιος είπε ήταν να αποτελέσει ένα αδερφάκι του MIT. Αν αντιστρέψουμε τη χρηματοδότηση όμως, ε, δηλαδή παίρνουμε τώρα δημόσια κονδύλια και τα διανέμε στην Ευρώπη, αυτό κάνει αυτό το Ινστιτούτο. Τώρα, χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, οι δεξιότητες των ερευνητών, ήταν ένα ερώτημα. Το θέμα δεν είναι ε, αν θα έχουμε περισσότερα χρήματα, αλλά αν θα τα διαθέσουμε στη σωστή θέση. Αδιάβασα πολλά άρθρα, μου λένε κάποιοι, ότι για να λύσεις προβλήματα δεν τους πετάς χρήματα. Μα αυτό θα κάνουμε τελικά. Και αφού δεν έχεις αρκετά χρήματα για να τα ρίξεις πάνω σε όλα τα προβλήματα, θα πρέπει να κάνεις ευφυείς επιλογές. Γιατί θεωρούν τόσο πολύπλοκες στις υποτροφίες, ίσως γιατί δεν είναι υποτροφίες ακριβώς, δεν, είναι επιδοτής ακριβώς, είναι και οι συμβάσεις που έχουν ε, ε, παραδοτέ αποτελέσματα και το 95% της χρηματοδότησης για τη βασική έρευνα προέρχεται από εθνικές πηγές και γι' αυτό εκεί πηγαίνουν και οι ερευνητές. Είναι πιο εύκολο από το να ζητήσουν ε, ευρωπαϊκή επιδότηση, ευρωπαϊκή υποτροφία. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα τελευταία. Τι άλλο να σχολιάσω. Όχι, θα σταματήσω εδώ. Thank you, Patrick. πολλά σχόλια ε, σχετικά με αυτά που είπες και ιδιαίτερα με την έννοια της αριστείας. Τώρα, βεβαίως, η αναζήτηση της αριστείας και η επιβράβευση της αριστείας οδηγεί σε δίκαια αποτελέσματα ή μήπω έχουμε κάποιες γεωγραφικές αδικίες εδώ. Και από εκεί και πέρα τα top πανεπιστήμια, τα καλύτερα πανεπιστήμια ε, και στον τομέα της έρευνας είναι καλύτερα και ξέρουν πώς να, πού να επενδύσουν κτλ. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Σαπίρ. Ο κύριος Όλμπριχτ αναφέρθηκε στην αισιοδοξία ή όχι για τη στρατηγικά γενικότερα. Θα απαντήσω στον κύριο Όλμπριχτ. Μετά θα αναφερθώ στο, ε, στη χρηματοδότηση στην Ευρώπη και μετά θα αναφερθώ στο τελευταίο ερώτημα για την αριστεία. Για την αισιοδοξία εσείς θα πρέπει να απαντήσετε, η πολιτική, όχι εγώ. Εσείς θα κάνετε τις επιλογές. Εμείς είμαστε εμπειρογνώμονες, αλλά δεν ήμουν σε θέση εγώ ως εμπειρογνώμονας να ξέρω κατά πόσο εσείς είστε σοβαροί ή όχι. Κάνετε απλώς δηλώσεις για, το, για την Ευρώπη 2020 ή διαθέτετε και τα χρήματα. Είστε σοβαροί. Εγώ δεν χρειάζεται να είμαι αισιόδοξο. Εγώ απλώ παρατηρητή είμαι και αναλύω την κατάσταση. Το υπήρχε η Σύνοδος Κορυφής ανεβλήθη από τον Οκτώβριο του Δεκέμβρη εξάνα ανεβλήθη σας όπως θα ξέρετε για το Φεβρουάριο έτσι εννοώ τη Σύνοδο Κορυφής για την καινοτομία καταλαβαίνω κατανοώ την ανάγκη για αναβολή και είναι ζωτική σημασία στο να γίνουν ορισμένα πράγματα για το ευρώ αλλά και η καινοτομία είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε είναι θέμα επι, επιβίωσης του ευρώ. Ναι, αλλά για την καινοτομία που είναι το μέλλον της Ευρώπης, αν δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον, ούτε η Ευρώπη θα επιβιώσει γενικότερα. Γι' αυτό είπα στην εισαγωγή μου ότι η ευρωπαϊκή κρίση είναι σοβαρό θέμα. και δεν μιλάμε για επιβίωση των επόμε... τους επόμενους μερικούς μήνες και μετά πράγματα θα γίνουν ε, ρόδινα. Όχι. Αντιθέτως βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο γενικότερα. Όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα δεν ε, ο κόσμος μας δεν πάει μοναχά από τις ανεπτυγμένες και οικονομίες, τις αναδιόμενες οικονομίες. Μιλάμε και για, αν θέλετε, γεωγραφική μετατόπιση από τη Δύση στην Ασία. Ε. Τέλος πάντων, για την αισιοδοξία επαναλαμβάνω δεν είναι δικό μου το θέμα. Είμαι στη διάθεσή σας, εσείς είστε οι εκλεγμένοι πολιτικοί και όχι εγώ. Δεύτερο ερώτημα, κατά πώς τα χρήματα εξοδεύονται με τον καλύτερο τρόπο στην Ευρώπη. Η απάντηση είναι δυστυχώς όχι. Όχι πάντα. Και η Μαρία Καβάγιο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω στο θέμα αυτό και όταν και όταν ήταν στην Πορτογαλία και όταν ήταν στην Κομισιόν και τώρα που είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι τα πράγματα από όλε τι οπτικέ γωνίε. Και αυτό που είπε είναι σωστό. Είναι τρομερό να βλέπει κανείς ότι ε, στους ερευνητές δεν αρέσουν τα προγράμματα. Τους αρέσει όμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Τι να πει κανείς. Έχει δίκιο λοιπόν η Μαρία Καρβάγιο η οποία τονίζει την ανάγκη για ένα καλύτερο σύστημα, λιγότερη γραφειοκρατία και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τι. Ε, μπορούμε να πάμε άλλο ένα βήμα μπροστά. Μήπως πρέπει να μεταρρυθμίσουμε και την Κομισιόν που διαχειρίζεται τα ποσά αυτά. Θεμητό νομίζω το ερώτημα. Αλλά εγώ θα ρωτήσω και κάτι τι άλλο. Μήπως πρέπει η ευθύνη αυτή να φύγει τελείως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πάει σε μια ανεξάρτητη αρχή. Εγώ προσωπικά θα ήμουν υπέρ μιας πραγματικής ανεξάρτητης υπηρεσίας. Πραγματικής όμως, όχι Μικη υπηρεσία, υπηρεσίας, πραγματικής Γιατί με, με δημοσιονομική αυτονομία, ε, όταν λέω πραγματική ανεξάρτητη αρχή λοιπόν για τα θέματα έρευνας και τεχνολογίας και καινοτομίας. Σας ρωτώ εσάς, είναι δική σας δουλειά αυτή. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν μπορώ και την ανάλυση να κάνω και τις αποφάσεις να παίρνω. Τρίτο θέμα τώρα. Ε, αριστεία ε, και συνοχή. Το ερώτημα είναι επίση πολύ θεμητό γιατί εμείς στην Ευρώπη είμαστε περήφανοι για την αλληλεγγύη και τη συνοχή και ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε στην οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε ε, ε, είναι ακόμη πιο σημαντική η, η συνοχή και η αλληλεγγύη. Δεν το υποτιμώ το ερώτημα και την ανάγκη γι' αυτό. Αλλά εφόσον μιλάμε εδώ για την έξυπνη ανάπτυξη, είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε και τεράστια σημασία του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τα ταλέντα και να τα προωθήσουμε και να προσελκύσουμε ταλέντα ίσως και απαλού. Και εδώ, γι' αυτό τον ανταγωνισμό μιλώ ανταγωνισμός για την αριστεία, για να βρούμε τα ταλέντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμελήσουμε τη συνοχή και την αλληλεγγύη. Απλώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλους μηχανισμούς. Τι κάναμε στο παρελθόν. Στο παρελθόν μπερδεύαμε την αριστεία και τη συνοχή και προσπαθούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε με ένα ενιαίο εργαλείο και έτσι δεν καταφέρναμε ούτε τόνο ούτε τ' άλλο. συμφωνώ για τους στόχους, αλλά με διακριτά εργαλεία, ε. Για αν με άλλο τρόπο θα επιλέξουμε και θα αγωνιστούμε για να επιτύχουμε την αριστεία και με άλλο τρόπο τη συνοχή. Ευχαριστώ Αντρέ. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της πρώτης συζήτησης. Να επανέλθω σε κάποια από τα θέματα τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια πριν κλείσω τη συζήτηση. Το πρώτο θέμα είναι ότι τώρα περνάτε σε μια συζήτηση εκ νέου για τον προϋπολογισμό. Όταν το Κοινοβούλιο συζητάει τον προϋπολογισμό ε, λέγει ότι ασχολείται ο προπολογισμό αποκλειστικά με θέματα τα οποία είναι αυτό που λέμε value for money. Δεν είναι δηλαδή ε, επενδύσεις οι οποίες μπορεί να πάνε ε, στράφη ούτε και μπορεί επίσης να δαπανηθούν χρήματα χωρίς έλεγχο. Έχουν έρθει στην επιφάνεια θέματα τα οποία αφορούν και το, πλαίσιο, το πρόγραμμα πλαίσιο 5 και 6 και ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθείται η επίδοση των προγραμμάτων αυτών είναι το ποσοστό της επίτευξης των στόχων και οι επιρροές, επιπτώσεις και συνέπειες που έχουν δυστυχώς τα προγράμματα αυτά δεν αξιολογείται ποτέ παρότι η προσπάθεια υπάρχει. Λοιπόν, τα προγράμματα πλαίσιο είναι, θα έλεγα, το μέσο με τα οποία τα προγράμματα τα οποία θα επιδιώξουμε πρέπει να είναι αηφόρα και έξυπνα. Αλλά θα πρέπει και η αξιολόγησή τους να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις και ε, τα αποτελέσματα γενικότερα των προγραμμάτων αυτών, του 7ου, του 8ου κτλ. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε και την εσωτερική διακυβέρνηση μεγάλων προγραμμάτων όπως το ΙΤΕΡ και τον Γαλιλαίο. Τα προβλήματα διακυβέρνησης τα οποία συνάντησα όταν τα ανέλησα είναι απίστευτου μεγέθους. Νομίζω ότι έχετε τα μεγαλύτερα ερευνητικά προγράμματα θα έλεγα στον κόσμο. Ε, το μόνο μεγαλύτερο από το ΙΤΕΡ είναι ο διαστημικός σταθμός αλλά στην ουσία τα προχωράτε τα προγράμματα αυτά χωρίς ένα δεδομένο μηχανισμό διακυβέρνησης και χωρίς σωστό συνδυασμό των συμμετεχόντων. Να λοιπόν τι μπορεί να κάνει ε, το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να αποτρέψει τα πράγματα για μια ακόμη φορά να πάνε άσχημα. Δεύτερη παρατήρηση. Εγώ είμαι ο παδός των ευθυνών ε, μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορεί κανείς να μεγαλώσει τον προϋπολογισμό. Και υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν σχετικά με, την, με τον ιδιωτικό τομέα και με τα κίνητρα που μπορεί να δώσει κανείς τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε κίνητρα στην μεταφορά τεχνολογίας ανάμεσα στα πανεπιστήμια και την βιομηχανία, είμαστε πίσω εδώ, Αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Ευρεσιτεχνία, αυτό ήταν θέμα συζήτησης εδώ και λίγα χρόνια, τώρα όμως σιγά σιγά το σκουπίζουμε κάτω από το χαλί. Δεν είναι μια ενιαία αυτόνομη λύση, αλλά είναι ένα κομμάτι από τις πιθανές λύσεις. Τέλος θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αλλάξουμε επίπεδο προς τα πάνω. Ε, το ακρόνιμο CATS e στα αγγλικά κομβικές ε, τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε, να βελτιωθούμε ποιες θα μας καταστήσουν ικανούς εν πάση περιπτώσει όχι μόνο να αποσβέσουμε τη συγκεκριμένη επένδυση αλλά να επηρεάσουμε πάρα πολύ θετικά και τον ευρύτερο οικονομικό τομέα σε σχέση με τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσει τύπης τουλάχιστον να επιδιώξει και να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετικά με τους δείκτες είναι πρώτον η διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών που ακολουθούνται η ανάγκη να δοθούν απαντήσεις στα κομβικά προβλήματα, πώς ανταποκρίνεται κανείς στην ικανοποίηση, για την ικανοποίηση των συγκεκριμένων δικτών, για την παρακολούθηση όλων των δικτών ανάπτυξης και για την ανάληψη της ευθύνης στην περίπτωση επίτευξης ή μη επίτευξης των στόχων. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στη Λισαβόνα και στο 2020 και αυτή η διαφορά θα πρέπει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η κατανομή των ευθυνών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι κάτι το οποίο είναι πλέον διακριτό ανάμεσα στις διάφορες γραμμές της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι σε τακτική βάση όλα αυτά είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε πώς επιτυγχάνονται στα πλαίσια της τραγικής του 2020 Νομίζω αυτό θα πρέπει να γίνει ήδη τον επόμενο χρόνο και όχι να περιμένουμε μια δεκαετία. Να ευχαριστήσω όσους πήραν μέρος στη συζήτηση, να ευχαριστήσω για όλα τα σχόλια τα οποία παρουσίασαν και τις ιδέες τους και να ευχηθώ σε όλους μια καλή συνέχεια στην ενδιαφέρουσα αυτή συζήτησή σας. Και ευχαριστώ την Χάουγκ επίση ε, για, ε, ε, για τον σωστό τρόπο με τον οποίο κατευθύνει τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ ολόκληρο το πάνελ και του, τους εμπειρογνώμονες. Βέβαια έχουμε λίγο ξεπεράσει το χρόνο, γι' αυτό ζητώ αλλαγή σκηνικού πάρα πάρα πολύ γρήγορα εδώ. Α, ah, thank you very much.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε αμέσως. Ο έχουμε το δεύτερο πάνελ τώρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αηφόρα ανάπτυξη. Ο στο οποίο λαμβάνει μέρο ο Κρίστιαν Ίγγενχόφερ από το Κέντρο Ευρωπαϊκών ε, Μελετών. Μετά έχουμε τον Βάλτερ Μπόλτς, αντιπρόεδρο από το και από το Συμβούλιο των ε, Ρυθμιστικών ε, Αρχών Ενέργειας. Μετά έχουμε τον Μύροσλαβ Τραϊκάς, από την Πολωνία, από την Ακαδημία Επιστημών και η moderator είναι η Ούλρικε Γκερό επικεφαλής του γραφείου του Βερολίνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Παρακαλώ. Η κυρία Γκερό, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τιμά ο ρόλος του moderator εδώ. Δεν είμαι ιδιαίτερη, ε, δεν είμαι η δημον για το Green New Deal. Δεν είμαι ιδιαίτερα γνώστη των θεμάτων της πράσινης αϊοφόρου ανάπτυξη γι' αυτό, αλλά ελπίζω να τα καταφέρω. Η ενέργεια είναι σημαντική και η επιλογή των μειγμάτων πολιτικής στον τομέα της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι η χώρα μου βρίσκεται στο κέντρο διαφόρων χωρών παραγωγών ενέργειας, διαμετα στον ενέργειες και τα λοιπά. Επίσης άρα έχουμε μια κάποια εμπειρία από όλα αυτά. Η ενέργεια επίσης είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει καθημερινά. Ε, ε η μεταφορά ενέργειας, αποτελεσματικότητα, ενέργειας, τιμή της ενέργειας είναι κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Ενδιαφέρονται λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολίτες για το θέμα ενέργειας, ε, έρχονται πιο κοντά ο ένας τον άλλον μέσω της ενέργειας. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε επίσης εμείς είναι το θέμα της πολιτικής και του μείγματος πολιτικής και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα πέντε λεφτά που έχω στη διάθεσή μου θα ήθελα να πω το εξή. Η ενέργεια είναι το επίκαιρο ή καυτή πατάτα του 21ου αιώνα. Πρέπει να αφιερώσουμε λοιπόν χρόνο και να σκεφτούμε για τις βιώσιμες ενέργειες. Και Ξαναλέω ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, της κατάρτισης αυτής και της πολιτικής ενέργειας της Ευρώπης. Ε, μπορεί η Ευρώπη, η Ευρώπη να έχει μια κοινή ενοποιημένη αγορά εργασίας. Υπάρχουν Επίσης, ε, πολλοί παράγοντες και παράμετροι που επηρεάζουν την ε, ε, τομή της ενέργειας της ενεργειακής υποδομής για τη δημιουργία δικτύων και τη δημιουργία νέων βιώσιμων δικτύων χρειάζεται τα αστρονομικά ποσά. Μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να τα καταφέρει. Τρίτο θέμα, η ενέργεια είναι κάτι όπου παίζουν σημαντικό ρόλο οι α, ε, εθνικές υποψίες. Ε, εγώ προέρχομαι από τη Γερμανία, από το Βερολίνο και πραγματικά ε, σας λέω ότι υπάρχουν υποψίες, θεωρίες ε, συνωμοσιών, ε, στρατιωτικών συνωμοσιών, πυρηνική ενέργεια δεν είναι πολύ αγαπητή στη Γερμανία. Σχετίζονται επίσης ε, τα θέματα ενέργειας με το περιβάλλον α, παίρνουμε, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και ένα καλό μείγμα πολιτικών στην ενέργεια. Επίσης τι θα γίνει στην οικονομία και πώς θα επηρεάσει αυτό το, ε, το, ε, θα προχωρούμε προς ευρωομόλογα ή όχι. Θα τολμούσα να πω ότι ο επόμενος προϋπολογισμός και το οικονομικό το, ο επόμενος προϋπολογισμός ή προϋπολογισμοί μάλλον ε, μετά το 2014 θα είναι ενδεχομένω έργα βιτρίνας απλώς και επί της ουσίας μπορεί να μην κάνουν τίποτα. Τολμώ να το πω, τολμώ να ρωτήσω. Λοιπόν, τους, τα μέλη του Πάνερ. Υπάρχει πιθανότητα να φτιάξουμε μια κοινή αγορά ενέργειας και ποιο κομμάτι θα καλύπτεται από την πράσινη ενέργεια, σε αυτή την κοινή ενέργεια. Μπορεί η αγορά να δώσει κατευθυντήριες γραμμές. Είχα στη διάθεσή μου δυο έγγραφα και κάπου διάβασα το εξής αριθμό για τις δαπάνες μεταφορών και ενέργειας το 99% είναι μη ευρωπαϊκό και το 1% μόνο είναι ευρωπαϊκό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Το μπορούμε να συνεχίσουμε με 99% εθνικές δαπάνες και 1% μόνο ευρωπαϊκή δαπάνη. Θα μπορούμε να αλλάξουμε, να τρέψουμε τα ποσοστά αυτά. αν μας χρειάζονται χρήματα για τον τομέα της ενέργειας, πώς μπορούμε να αποδεσμεύσουμε ποσά από άλλους τομείς και να τα φέρουμε στην ενέργεια. Πώς μπορούμε να πάρουμε χρήματα από πολιτικές όπως η κοινή αγροτική πολιτική ας πούμε που θεωρούνται πολιτικές συνοχές ή άλλες πολιτικές συνοχές μπορούμε να το κάνουμε αυτό Πιστεύω ότι η ενέργεια είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα των επόμενων της επόμενης δεκαετίας και δίνω το λόγο του κύριο Μπόλτς ο οποίος είναι αντιπρόεδρος στην Υπηρεσία για τη Συνεργασία Εθνικών Ενεργειακών Ρυθμών, ε, Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, για την αηφόρο ανάπτυξη, μια και εκπροσωπώ τις ρυθμιστικές αρχές για την ενέργεια, θα αναφερθώ στα θέματα της ενέργειας αποκλειστικά. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τους στόχους των προγραμμάτων για την Ευρώπη του 2020 για ανταγωνιστική και πράσινη και αηφόρο οικονομία. Όπως είπαμε, το πρώτο κομμάτι, οι στόχοι της Λισαβόνας δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά πετύχαμε. Και τώρα για δεύτερη φορά θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε κάπως την απόδοσή σας, την απόδοσή μας μάλλον, και να δούμε αν μπορούμε να καλύψουμε τον σκόπελο που αντιπροσωπεύει η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία βέβαια γίνεται όλο και πιο ακριβή και θα δούμε πόσα χρήματα περισσεύουν για τον καταναλωτή να δαπανίσει σε άλλους τομείς, ταυτόχρονα καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες του καταναλωτή. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι τους οποίους θα πρέπει να πετύχουμε. Καταρχάς θα πρέπει να καταστήσουμε λειτουργική την εσωτερική αγορά. Έχουμε προχωρήσει στην απελευθέρωση της αγοράς τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχουμε κάνει κάποια βήματα προόδου, αλλά νομίζω ότι το τρίτο πακέτο, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον επόμενο χρόνο, θα συνεισφέρει κατά πολύ έτσι ώστε οι αγορές ενέργειας να φτάσουν σε μια φάση όπου να είναι πράγματι αποτελεσματική, να έχουμε επίσης τιμές ενέργειας που να ορίζονται από την αγορά, και να λειτουργούν οι αγορές της ενέργειας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να απορροφούν τις προστιθέμενες αξίες των εφαρμοζόμενων πολιτικών για την ανανέωση των ποιών ενέργειας και έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε αποτελεσματικότεροι και σε άλλους τομείς όπως η κατοικία κτλ. Ε, βάζουμε επίσης και την κάλυψη κάποιων αναγκών καθολικού ενδιαφέροντος κοινή ωφέλεια όπως τα λέγαμε στα πλαίσια της αγοράς ενέργειας και θα πρέπει οι αγορές ενέργειας να λειτουργούν σωστά, δίκαια και παρά όλα αυτά τα επιπλέον κόστη σε εισαγωγικά. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι επίσης ότι όλα τα συστατικά για την λειτουργική αγορά της ενέργειας να είναι στη θέση που πρέπει δηλαδή η πολιτική ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέες τεχνολογίες, ενίσχυση των δυνατοτήτων των καταναλωτών και εξωτερική διάσταση της προμήθειας ενέργειας. Θα στρέψω την προσοχή μου κυρίως στο πώς εμείς μπορούμε να καταστήσουμε τις υποδομές να δουλέψουν καλύτερα και πώς ακριβώς οι υποδομές και κυρίως οι δικτυωσεις θα παίξουν τον ρόλο που καλούνται να παίξουν. Είμαστε στα πλαίσια μιας διαδικασίας να πετύχουμε τους στόχους αηφορίας και περιβάλλοντος που είχαμε θέσει. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πλήρως τον τομέα της ενέργειας. Ήδη το 2015 μετά από μακρές επενδύσεις θα πρέπει να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς καμία εκπομπή καυσαερίου του άνθρακα. Σήμερα η δημιουργία ηλεκτρισμού ε, είναι ένα μείζον παράγων εκπομπών και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Συνεπώς εμείς θα περάσουμε σε κάτι λιγότερο από τα δύο τρίτα της ενέργειας που θα παραμείνουν βέβαια σε, ε, που θα παραμείνει η παραγωγή τους σε ορυκτά καύσιμα σε δίκτυα επίσης ε, τα οποία θα είναι απαραίτητα για την κάλυψη των περιφερειακών αναγκών στην Ευρώπη. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε αρκετά χρήματα. Το σύνολο των ποσών είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα υπολογίσει κανείς γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια και πολλά πρότυπα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες των επενδυτών, αλλά τεχνικά υπάρχει μια ανάγκη επενδυτική για τις υποδομές, ιδιαίτερα στον τομέα του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού. Το θέμα είναι πώς θα τα ορίσουμε αυτά, ποια θα καλυφθούν από το εθνικό, εθνικό επίπεδο, ποια από το ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια θα καλύψουν οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της Ένωσης και σε ποιες φάσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν επίσης και κάποιες βασικές αρχές τις οποίες θα πρέπει να βασίσουμε στις εμπειρίες που είχαμε με διάφορες προηγούμενες πολιτικές που χρησιμοποιούσαμε στην Ευρώπη σε διαφορετικές συνθήκες. Ποια είναι τα βασικά μαθήματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε. Πρώτον, είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε τις αγορές ε, σαν τους, τις βασικές πηγές επένδυσης. Η πολιτική δεν είναι πάρα πολύ καλή στη βέλτιστη χρήση των επενδυτικών διαθεσίμων. Η Γερμανία είναι ένα καλό παράδειγμα που τώρα συνειδητοποιούν ότι η πολιτική που προκάλεσε τις επενδύσεις για τη φωτοβολταϊκή ενέργεια έχει φτάσει σε κάποια επίπεδα κόστους που είναι πλέον ανυπόφορα. Είναι πολύ υψηλά. Δεν είμαστε λοιπόν σε μία περίοδο αποκλειστικά της πολιτικής να ορίζει τις υψηλές επενδύσεις και να προσπαθεί να τις καλύψει. Πρέπει λοιπόν εμείς να εμπλέξουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους ιδιώτες της αγοράς και οι μοναδικές αλλαγές τις οποίες θέλουμε εμείς ουσιαστικά να κάνουμε είναι να ευνηγραμμίσουμε τις πολιτικές αυτές με τους στόχους που έχουμε στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερον, θα πρέπει να διαρρυθμίσουμε τα διακανονιστικά πλαίσια σταδιακά, να υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος χρόνος έτσι ώστε να δώσουμε στην αγορά τη δυνατότητα να αποσβέσει την επένδυση και να υπάρξει και η απαιτούμενη ασφάλεια για τις επενδύσεις αυτές ε, για τις νέες μορφές ε, δικτύων αποδοτικότητας κτλ. Και εδώ η Γερμανίδα ε, χρησιμοποιώ πολλά γερμανικά παραδείγματα βέβαια, αλλά αν η γερμανική πολιτική λέγει ότι θα πρέπει να βγούμε από την πυρηνική ενέργεια και να περάσουμε στο φυσικό αέριο. Τώρα έχει 20 μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλήρως. Υπάρχει ένας κίνδυνος λοιπόν οι πολύ μεγάλες πολιτικές επενδυτικές αποφάσεις να λαμβάνουν χώρα μεν, αλλά μετά κάποιες επιμέρους αλλαγές να καθιστούν αυτές τις πολιτικές ανεφάρμοστες. Και εδώ η εναρμόνιση των ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σημασία, η ε, πολιτική ενέργεια όσο γίνεται πιο ευρωπαϊκή θα εξαρτάται από τα ευρωπαϊκά κόστη και απαιτείται εναρμονισμένη αντιμετώπιση. Υπάρχει εδώ συγκεκριμένος ρόλος και για ευρωπαϊκές επενδύσεις κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Οι ικανότητες, οι επενδυτικές, οι ευρωπαϊκές είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με αυτά που απαιτούνται. Αλλά οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοδότησης μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο όταν οι εθνικές επενδύσεις δεν είναι εφικτές γιατί το κόστος και όφελος είναι θα έλεγα κάτι το οποίο κατανέμεται ανάμεσα σε διάφορα χώρες. Αν δηλαδή το κόστος το καλύπτει κανονικά μία χώρα αλλά το όφελος τον έμεται μία άλλη χώρα, σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατανομή του κόστους και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει τις επενδύσεις οι οποίες σε εθνικό επίπεδο είναι δύσκολες. Μηχανισμοί απόδοσης κινήτρων. Είναι προτιμότερη από την πλήρη χρηματοδότηση την ευρωπαϊκή που έτσι και αλλιώς είναι no-go επιλογή λόγω της έλλειψης διαθεσίμων επενδύσεων. Το θέμα είναι πώς μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες χρηματοδοτικούς μηχανισμούς όπως το Ταμείο Συνοχής κτλ. Και, και να μην δημιουργήσουμε κάτι το εντελώς ξεχωριστό. Δεν μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Τα ευρωπαϊκά όργανα δεν ήταν πάρα πολύ ικανά για τη διαχείριση των ε, χρημάτων αυτών, όπου έχουν δοθεί τέτοια χρήματα, απεδείχθη ότι ήταν πολύ συγκεντρωτική η ισορροπία η οποία διασφαλίστηκε για την κατανομή των χρημάτων και δεν υπήρξε συγκεκριμένη προσοχή σε κάποια προγράμματα και υπήρξε κατανομή και πολυδιάσπαση και ακριβώς λόγω των μικρών ποσών που κατέληξαν τελικά δεν υπήρξε η απαιτούμενη αποτελεσματικότητα. Απαιτείται λοιπόν να δούμε τι νέα προγράμματα μπορούμε να βρούμε και γι' αυτό θα απαιτηθούν κάποια χρόνια. Πέραν της χρηματοδότησης υπάρχει το θέμα της ελάττωσης των κινδύνων, η κοινωνικοποίηση των κινδύνων. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει την σύλληψη σε εισαγωγικά ενός προϋπολογισμού. Ευχαριστώ κύριε. Δεν ακολούθησα τη σωστή σειρά. Νομίζω ότι καλό θα είναι να ακολουθήσουν τώρα ο Μύρος Λαβδρούγκας της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών. Ακριβώς επειδή προέρχεστε από μια διαφορετική πραγματικότητα, μια χώρα στις οποίες οι πολιτικές της Γεωργίας σαν παράδειγμα είναι πολύ σημαντικές και γι' αυτό μετά θα περάσουμε στον Κρίστιαν Ιγενχόφερ ο οποίος ασχολείται για το κλίμα, με το κλίμα και την ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως είμαι ο μόνος που θα μιλήσω από ένα πρίσμα διαφορετικό, το πρίσμα της γεωργίας. Η στρατηγική 2020 είναι ιδιαίτερη σε ό,τι αφορά ε, τη γεωργία, γιατί σχετίζεται με την ασφάλεια των τροφίμων. Λόγω της παγκόσμιας κατάστασης, ε, ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα. Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με τις χώρες Μερκοσούρ και από αυτές τις διαπραγματεύσεις υπάρχουν φόβοι αλλά και απειλές. Ε, Απειλείται ουσιαστικά και το μέλλον του γεωργικού τομέα στην Ευρώπη. Η γεωργία σχετίζεται στενά βέβαια με τα ενεργειακά ζητήματα. Σήμερα αντιμετωπίζει δυσκολίες. Υπάρχουν ολόκληρες εταιρείε και κοινωνίες που δεν είναι ευαισθητοποιημένες ε, στον ε, για τον τομέα της γεωργίας, δεν καταλαβαίνουν ε, γιατί δίνονται ενισχύσεις στους αγρότες. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται σε ένα κατώτατο επίπεδο ε, η πρακτική αυτή να συνεχιστεί αν θέλουμε να επιτύχουμε τους μελλοντικού στόχους. Δεν θα πρέπει βέβαια να επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα, να σας αιτιολογήσω όλα αυτά, αλλά θα αναφέρω κάποιους παράγοντες. Πρώτα απ' όλα στην Πολωνία Λέμε πολλές φορές ότι η κοινή γεωργική πολιτική χρησιμεύει μόνο στο να γεμίζουν οι τσέπε των αγροτών. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εμείς οι κοινοτικοί καταναλωτές έχουμε πιο φθηνά τρόφιμα χάρη στην κοινή γεωργική πολιτική. στο πλαίσιο και της κανονικής διαδικασίας ανταγωνισμού. Επίσης, η ΚΑΠ βοηθάει να δοθεί μεγαλύτερο, μεγαλύτερο δυναμικό και σε άλλους τομείς. Σε ό,τι αφορά την Πολωνία, το 90-95% των κονδυλίων της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής δαπανώνται για την αγορά διαφόρων αγαθών που προέρχονται από άλλους τομείς. Υπάρχει λοιπόν ένας δυναμισμός, ε, υπάρχει νέα όθηση στην οικονομική ανάπτυξη για άλλους τομείς, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ενεργειακά ζητήματα, θα επανέλθω. Νομίζω ότι η κοινή γεωρική πολιτική σήμερα είναι παρκώ όρημη, έχει φτάσει στη στιγμή δηλαδή όπου πρέπει να τεθεί ε, ένα ερώτημα ακόμη και για τον τίτλο. Δηλαδή νομίζω ότι θα έπρεπε να αλλάξει τίτλο, να ονομάζεται δημόσια πολιτική τροφίμων και αγαθών, γιατί υπάρχει το θέμα της ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όλα αυτά που είναι συναφή με αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό λοιπόν ζήτημα. Εγώ αναγνωρίζω την προστέμενη αξία της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατεύθυνση, τον προσανατολισμό που έχει, να έχουμε δηλαδή παραγωγή ποιοτικών τροφίμων, υγιών τροφίμων. Γι' αυτό έχουμε και τέτοια τρόφιμα, άλλωστε ποιοτικά και υγιεινά τρόφιμα και αυτό σίγουρα επηρεάζει και την υγεία των κοινωνιών τη δημόσια υγεία. Και βέβαια μακροπρόθεσμα επιτρέπει και τη μείωση του κόστους ε, που θα πρέπει να απομιστούν ε, τα κοινωνικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι αφορά τώρα τη διασύνδεση της κοινή γεωργικής πολιτικής και της γεωργίας εν γέννη με τα ενεργειακά ζητήματα. Νομίζω έγινε λόγος ε, και στο πρώτο πάνελ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την καινοτομία. Η καινοτομία η οποία σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο και με τη μείωση της παραγωγικότητας. Είπαμε ότι θα πρέπει να γίνεται επιλογή των σχεδίων με βάση τον ανταγωνισμό. Κατά την προσωπική μου άποψη υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει την γεωργία παντού στον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το ενδεχόμενο θέσπισης αυτού του νέου μέσου για την παροχή γεωργικών τεχνολογιών ε, με την ε, χαμηλότερη δυνατή τιμή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε ότι οι νέε τεχνολογίε, οι πιο καινοτόμε τεχνολογίε είναι πολύ δαπανηρέ. Και γι' αυτό ε, δυσκολεύονται να τι αποκτήσουν ορισμένοι αγρότε. Νομίζω λοιπόν ότι η καινούργια πολιτική θα μπορούσε να διαθέσει πόρου υπέρ τη ανάπτυξη, περνώντα ακριβώ μέσα από αυτό το εργαλείο. Επίση, υπάρχει και το ζήτημα τη ανταγωνιστικότητα. ιδίως ό,τι αφορά τις ε, καλλιέργειες για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Πιστεύω ότι η παραγωγή τροφίμων ή τα γεωργικά προϊόντα πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προορίζονται για τη διατροφή. Η γεωργική παραγωγή πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο 70% της ε, ζήτησης τροφίμων στην Ευρώπη. Λένε όμως κάποιοι ότι είναι τόσο πλούσια η Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να αγοράζει τα πάντα ε, παντού και με την τιμή που θέλει. Αυτό θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε ανταγωνισμός, αν δεν υπήρχε πραγματικός ανταγωνισμός αλλά πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ε, την αγορά ζάχαρης, για παράδειγμα. Η Πολωνία ήταν ε, εξαγωγέα ζάχαρης. Οι λιανικές τιμές σήμερα όμως είναι πάρα πολύ υψηλές, ο υψηλότερο θα έλεγα επίπεδο εδώ και 30 χρόνια. Άρα δεν αληθεύει αυτό. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και να αρχίσουμε τις προτεραιότητες μας για το μέλλον. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, άκουσα όλα αυτά που είπατε. Έχουμε τις παραδοσιακές παλές πολιτικές και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τις εξυγχρονίσουμε και είπατε εσεί να τους αλλάξουμε και όνομα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Να δώσω τώρα το λόγο στον Κρίστιαν Ίγκενχόφερ που είναι Senior Research Fellow στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών Μελετών. Συγγνώμη που θα σας απογοητεύσω, δεν είμαι ειδικό για θέματα ενεργειακής, πολιτικής ενέργειας, αλλά είμαι ειδικό για το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα για την κλιματική αλλαγή. Τα πράγματα είναι απλά, τουλάχιστον θεωρητικά. Άμα κοστολογείς κανείς τον άνθρακα, μετά προχωρούν τα πράγματα και διοχετεύονται σε μέσω όλης της διαδικασίας και φτάνουμε τελικά σε ένα κάποιο νούμερο. Τα ξέρετε όλα αυτά, τα λέω όμως γιατί ε, αν το σύστημα το οικονομικό δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ απλό αυτό για σας αλλά το ξαναλέω αν δεν είμαστε αποτελεσματικοί αν δεν έχουμε ένα κάποιο καλό αποτελεσματικό οικονομικό σύστημα δεν μπορούμε να ε, πετύχουμε πολλά και βεβαίως ακούστηκαν διάφορα για τις αποτυχίες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά το πρόβλημα δεν είναι η, για την έρευνα και την ανάπτυξη το κομμάτι του δημοσίου αλλά το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα. Το ερώτημα είναι αν ανατρέψουμε τα ισχύοντα ποσοστά ή προστε... αυξήσουμε το μερίδιο του δημοσίου τομέα, αν τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει το ανα, ακούστηκε η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, για διαφορετικές υποδομές και τα και άκουσα με μεγάλη χαρά αυτά που είπε ο κ. Μπόλτς για το πως φαντάζεται να εξελίσσονται στο μέλλον τα συστήματα αυτά τα υποδομών συμπεριλαμβανομένες και τις γεωργίας και τα Αλλά Πέρα από όλα αυτά η στρατηγική 2020 περιλαμβάνει και το ο, θέμα της αποτελεσματικότητας των πόρων. Βεβαίω η αποτελεσματικότητα των πόρων πολλές φορές εξαρτάται από την τιμή των βασικών προϊόντων. μπορεί κανείς να επέμβει εκεί, να έχει εισαγωγή, φόρους κατά την εισαγωγή, φόρους κατά την εξαγωγή κτλ. Αλλά άμα τα σκεφτούμε όλα αυτά φτάνουμε πολύ γρήγορα στο στοιχείο ανταγωνιστικότητα όπου τα πράγματα αλλάζουν. Για να μην περιπλέξω ακόμη περισσότερο τα πράγματα θα ήθελα να πω ότι η στρατηγική του 2020 κατά την άποψή μου μοιάζει με μια δήλωση προθέσεων ή αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην το λέμε όμως σχέδιο και πρόγραμμα. Ε, δεν είναι τα πράγματα τόσο ο, σαφή. Τώρα ετέθη βέβαια και το θέμα του προεπλογισμού για, για την Ευρωπαϊκή Ένωση η πολιτική καθοδήγηση του προϋπολογισμού είναι σημαντική. Δημιουργεί ο προϋπολογισμός με άλλα λόγια κάποια κίνητρα, δίνει κάποια κίνητρα και προσελκύει επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Ε, είναι σημαντικό αυτό λοιπόν και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κάπου κατευθύνει. Βεβαίως από εκεί πέρα υπάρχει και ένα στοιχείο αλληλεγγύη στον προπολογισμό. Προσπαθεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι δυνατόν, να εξισορροπήσει κάποιες ανισότητες ή, εν περιπτώσει, να μοιράσει δίκαια το βάρος ή κάπως πιο δίκαια το βάρος. Από εκεί πέρα συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Σαπίρ, ότι ο προεπολογισμός πρέπει να προωθεί και την αριστεία. Αλλά ένα μεγάλο κράτος μέλος όπως η Γερμανία και η Γαλλία χρειάζονται τα μεγάλα κράτη-μέλη κοινοτικά κονδύλια για να προωθήσουν την αριστεία. Εγώ θεωρώ πως όχι. Θα μπορούσαν μόνες τους οι μεγάλες χώρες να το κάνουν αυτό. Άλλοι χρειάζονται τα κοινοτικά κονδύλια. Τέλος πάντων για να μην καθυστερώ ως Γερμανός προσπαθώ να μην καθυστερώ ε, τι μπορούμε συγκεκριμένα να κάνουμε εταιρική σχέση επενδύσεις τι, που θα έκανα τις επενδύσεις μου στις βαλτικές χώρες πρώτα πρώτα για την ενέργεια γιατί η υποδομή τους γυράσκει αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να ανανεώσουν να περάσουν σε μια νέα φάση και μπορούν κατευθείαν να πάνε στις νέες υποδομές από εκεί και πέρα ε, ε, αστικά κέντρα είναι πολύ σημαντικό να γίνουν επενδύσεις και εκεί θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα αστικά κέντρα τρίτο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε πέρα από τον προπολογισμό της Ένωσης να συμμετάσχουν σε, στην ενέργεια και άλλοι φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κτλ. Και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει και το ε, δίκτυο, το εσωτερικό, η κοινή αγορά κτλ. Εγώ τώρα για να απαντήσω μια ερώτηση που ετέθη στο προηγούμενο πάνελ για το Πού θα βάζα το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Θα το βάζα σε εταιρικές σχέσεις, εταιρικές συμβάσεις, στη, σε αστικά κέντρα. Εκεί νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ε, η κυρία Γκερό Η κυρία Χάουγκ ε, έχει το λόγο και πάλι. Ναι, λέει η κυρία Χάουγκ, έχω δύο ομιλητέ που θα ήθελαν το λόγο. Ο κύριος Πόλσεν. Η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ καλή, είναι εξαιρετική. Και αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να κάνω είναι να έχουμε μια ανατροφοδότηση για την ευρωπαϊκή προοπτική. Εμείς που καθόμαστε εδώ ενώ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως έχουμε μια καλύτερη προοπτική όταν προσπαθούμε να αποκομίσουμε μια ρεαλιστική εικόνα της κατάστασης. Ακούσαμε να γίνεται λόγος για την αλλαγή του κλίματος, το πρόβλημα της γεωργίας, το ρόλο της έρευνας. Ακούσαμε να γίνεται λόγος για την ενέργεια. Πέραν του κλίματος, Νομίζω ότι υπάρχει και ένα άλλο τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Άλλα ε, ε, νητρικά, άλλα τα φωσφορικά, άλλα τα και άλλα χημικά μολύνουν την, το έδαφος και για να βιοποκοδομηθούν χρειάζονται 500 χρόνια και το ίδιο συμβαίνει και στη θάλασσα. Ρίχνουμε στη θάλασσα πράγματα που μπορεί να μην βιοποικοδομηθούν ε, στο προβλέψιμο μέλλον. Μπορούμε να ξεκινήσουμε όμως με τον τομέα της γεωργίας. Είναι και τομέας που με ενδιαφέρει και εργάζομαι. Έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό για να αποτρέψουμε την αλλαγή του κλίματος. Θα μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε το διοξίδιο του άνθρακα εάν δεν οργώναμε. Αν δεν οργώναμε θα είχαμε ένα τεράστιο πλεόνασμα για πολλά χρόνια και θα μπορούσε να ισορροπήσει κάπως ε, ο πλανήτης Γη. Ε, θα πρέπει όμως να δούμε το εξής. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα αγριόχορτα και τα ζυζάνια όταν δεν οργώνουμε το έδαφος. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι ένα μεγάλο θέμα και θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε και πολλά χρήματα για να το λύσουμε. Βέβαια έχουμε τεχνολογία ε, που γνωρίζουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γνωρίζουμε ότι είναι και σε προσιτή τιμή. Η δασοκομεία, η γεωργική δασοκομεία θα μπορούσε να είναι απόλυτα αυτάρκηση σε ό,τι αφορά την ενέργεια. και η γεωργία θα μπορούσε να παράγει τρόφιμα χωρίς να μειωθεί παρά κατά το ελάχιστο δυνατότητά της αυτή. Έχουμε 6,7 δις άτομα στον πλανήτη και στο προβλέψιμο μέλλον θα φτάσουν τα 9 δις. Άρα, ό,τι έδαφος υπάρχει που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τροφίμων θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Και έχουμε και τον κύκλο ζωής ε, των ε, χημικών αυτών που σας είπα πριν. Μπορούμε γενικά να εξοικονομήσουμε ενέργεια εάν η γεωργία προσανατολιστεί προς το μέλλον και μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια. Θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο γενικά και έτσι με ένα για να δούμε πού είναι οι λεπτομέρειες που θα πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Thank you, I would like to come back to the... Ευχαριστώ, Ούτα. Θα ήθελα να επανέλθω στο στρατηγικό στόχο αυτού του πάνελ. Τι συζητάμε, τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και πιο που να χρησιμοποιεί καλύτερα τους πόρους που έχει. Η Κίνα από ό,τι ξέρω είναι πρωταγωνίστρια στην αιωλική ενέργεια. Χάσαμε την πρωτιά αυτή εμείς στην Ευρώπη. Γιατί, διότι χάσαμε την πρωτοπορία, τη τεχνολογική. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Πρέπει να φροντίσουμε να διατηρούμε την πρωτοπορία, την τεχνολογική σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, για να μπορούμε να επηρεάσουμε και το μέλλον. Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Έγκενχόφερ είπε ότι νομίζεις ότι η στρατηγική του 2020 είναι δήλωση προθέσεων και ε, αποστολής αλλά όχι συγκεκριμένο σχέδιο. Ίσως δεν κατάλαβα αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ακόμη κι αν δεν είναι συγκεκριμένο σχέδιο η στρατηγική 2020 πρέπει να βιαστούμε. Ε, ήδη αποτύχαμε μία διαφορά. Τώρα πρέπει να αναλάβουμε την πολιτική δέσμευση να κάνουμε κάποια πράγματα. Διαφορετικά θα αποτύχουμε και πάλι. Άρα οι αγορές, ο ιδιωτικός τομέας, ε, ο δημόσιος τομέας, τα κράτη-μέλη και η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστούν για να πάμε παρακάτω. Μετά μίλησες για την πολιτική καθοδήγηση, αν θες, που δίνει ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμό κατευθύνες γραμμές που μπορεί και χαρά αλλάζει. Είναι πιο σημαντικό αυτό, είπε, από το συγκεκριμένο μέγεθο των κονδυλίων. Πράγματι, τα κονδύλια της προ... του προπολογισμού του ευρωπαϊκού δεν είναι μεγάλα. Άρα, ναι, έχει δίκιο. Απλώ χαράσει κατευθυντήριε γραμμέ ο προπολογισμό. Αλλά εγώ ρωτώ τότε, μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Γιατί αυτό που είπες εσύ σημαίνει ουσιαστικά ότι κάποια κράτη-μέλη, αυτό που είπες εσύ μάλλον, ότι κάποια κράτη, μεγάλα κράτη-μέλη μπορούν κάποια πράγματα να τα κάνουν από μόνοι τους και δεν χρειάζονται κοινωτικά κονδύλια, τότε τι να πω. Η Γαλλία και η Γερμανία μπορούν να συνεχίσουν μόνοι τους. Μα δεν πρόκειται για κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση τότε και κατά τη δική μου, άποψη για να είμαστε επιτυχεί στο μέλλον θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί, να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Θέλω να πω ότι σε αυτά που είπε ο κύριος Έγκενχόφερ εδώ, εγώ δεν να υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. José Eu vou ser muito. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Μία ερώτηση η οποία νομίζω είναι αρκετά απλή. Η αηφόρος ανάπτυξη είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους πόρους. Μιλήσαμε επίσης και για τον φόρο που θα προέλθει από το διοξίδιο του άνθρακα και από το φόρο για την ενέργεια πιθανώς. Και εδώ είναι το ερώτημα και στρέφομαι στο σύνολο των ομιλητών. Μήπως ακριβώς η αγορά, α, τα έσοδα της αγοράς αυτής ε, που θα προέλθει από το διοξίδιο του άνθρακα να θεωρηθεί ε, σαν τμήμα των κοινοτικών ιδίων πόρων και να μην γίνεται αντικείμενο διαχείρισης από τα κράτη-μέλη. Και το ίδιο να ισχύσει και για τον φόρο για την ενέργεια που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ε, και στο περιβάλλον. Λοιπόν, ε, πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να ισχύσει. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι νέοι αυτοί πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αηφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σικεύσκη. Τα τελευταία χρόνια Προσπαθήσαμε να δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα της λειτουργίας των αγορών. Μας έδωσαν την εντύπωση ότι υπήρχε μια άγνοια σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι αγορές αυτές. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε με την αγορά της ενέργειας. Η αγορά της ενέργειας έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια της υπήρου μας και με πάρα πολλά πολιτικά ερωτήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει έλθει στην επιφάνεια πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Μπορούμε να έχουμε επανάληψη των φαινομένων που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια και σε άλλους τομείς, σαν παράδειγμα στον τομέα των πρώτων υλών για τα τρόφιμα. Πολλοί λένε δεν υπάρχει λόγος παραγωγής, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής. Αλλά αυτό εδώ δεν αγνοεί μήπως το θέμα της ασφάλειας των προμηθειών και πιθανές απειλές που μπορεί να δημιουργηθούν στο επίπεδο της προμήθειας σε τρόφιμα. Γιατί θυμίζω ότι η ασφάλεια στον τομέα της προμήθειας των τροφίμων είναι ίσως πιο σημαντική από την αντίστοιχη στον τομέα της ενέργειας. Πρέπει λοιπόν οι πολιτικοί να μπορέσουν να δουν σε ποιο βαθμό ε, και ποιον βαθμό μάλλον εξάρτησης μπορούν να δεχθούν στον τομέα των τροφίμων. Η Ευρώπη δημιούργησε την ΚΑΠ αμέσω μετά τον πόλεμο, μια περίοδο, περίοδο η οποία δεν ήταν και πάρα πολύ μακρινή χρονικά, για να αντιμετωπιστεί η πείνα που σοβούσε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο την εποχή. Λοιπόν, τίθεται εδώ το θέμα να προσπαθήσουμε να δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορέσει κανείς να ρυθμίσει τις αγορές. Και αυτό αφορά την ενέργεια και τις χρηματαγορές επίσης και το κόστος φυσικά να καλύψει κανείς όλα αυτά. Η πολιτική, εν πάση περιπτώσει, συνοχής επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μια αναπτυξιακή πολιτική. Και η κοινή αγροτική πολιτική παρέχει ένα επίπεδο ασφάλειας και στον τομέα των τροφίμικων αλλά και στον τομέα της υγιεινής των τροφίμων κυρίως και στο περιβάλλον. Το είπε άλλωστε και ο κύριος Δρούγας Συνεπώς ε, πρόκειται για κάτι το οποίο θα χαρακτήριζα δημόσιο αγαθό. Πώς μπορούμε να τα αξιολογήσουμε όλα αυτά στον συγκεκριμένο τομέα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο τομέα θα επηρεάσει τη συνοχή. Νομίζω ότι θα πρέπει και η εταιρική σχέση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να γίνει πραγματικότητα. Και υπάρχει γενικά εδώ το θέμα έτσι και αλλιώ τη αηφορία στην ανάπτυξη. Μιλάμε για την ενέργεια, αλλά σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για άλλα πράγματα. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να τα αναπτύξω όλα αυτά, αλλά Ε, πρέπει να δούμε και κάποια θέματα που συνδέονται με τη γεωργία και το περιβάλλον όπως η υδάτινη πόρη. Τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει πολύ το νερό όπως ίσως και η ενέργεια σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σχολιάσω αυτά που ανεφέρθη όλα αυτά που ελέγχθησαν από τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν συγκεκριμένη θέση ε, για ορισμένα πράγματα διότι πάντα υπάρχει και υπάρχουν και τα μεν και τα δε. Εμάς περιπτώσει σπούδασα και εγώ οικονομία και αγροτική οικονομία και αν δεν ξέχασα αυτά που μαθαίναμε τότε στο Πανεπιστήμιο νομίζω ότι η τιμή των σιτηρών ήταν το κεντρικό σημείο αναφοράς ε, στην αγροτική οικονομία. Τα πράγματα άλλαξαν βεβαίω τότε. Ε, τότε υπάρχουν καινούργιες σχέσεις, υπάρχουν καινούργιες εξαρτήσεις και εγώ δεν λέω ότι αμφισβητώ ότι θα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αμφισβητήσουμε την παραγωγή τροφίμων ε, από τους γεωργούς, από τους αγρότες αλλά υπάρχουν την σήμερα ημέρα και τεχνολογίες που μας ε, βοηθούν να έχουμε ό,τι τρόφιμο χρειαζόμαστε σε περίπτωση σπάνιδος ή σε περίπτωση εξαιρετικών συνθήκων. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να ερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες η, ο ανταγωνισμός η αύξηση παραγωγικότητας ε, είναι παράμετροι που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και οι οποίοι ε, αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από άλλα πράγματα ή έχουν βέβαια διαφορετική, την διαφορετική τιμή ε, δια, την πληρω, πληρώνουμε διαφορετικά για αυτά την σήμερα ημέρα να πω ότι στο παρελθόν οπότε τι ρόλο παίζουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ο προπολογισμό σε αυτή την όλη τη συλλογιστική σίγουρα μάθαμε από το παρελθόν ότι κάναμε λάθη, ότι αποτύχαμε γιατί υποτιμήσαμε την, το κόστος κάποιων μεταρρυθμίσεων και ε, αυτά όλα τα λάθη δεν θα πρέπει να τα ξανακάνουμε άρα μπορώ να φανταστώ ε, να χρειάζεται να επηρεάζει πολύ σημαντικά ο προπολογισμό στο μέλλον της Ευρώπης Ευχαριστώ. Είμαι παρατηρήτρια αυτή της ε, συζήτησης ουσιαστικά. Ξεκινήσαμε για το ε, πρασίνισμα και περάσαμε σε τέτοιες διαφορετικά θέματα. Βλέπω λοιπόν πόσο δύσκολο είναι κανείς να διαμορφώσει πολιτικές και να πάει από κάποιες παλιές σε κάποιες νέες πολιτικές. Αυτά έτσι απλά ως προβληματισμό. Θα επανέλθω αντίστροφα στο πάνελ. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Έγγενχόφερ, ε, μετά Ντρούκας, μετά Μπόλτσα αλλά να ξαναπώ αυτό το οποίο εγώ θα περίμενα ίσως ως απάντηση, γιατί κάποια από τα ερωτήματα νομίζω ότι πιο πολύ πηγαίνουν ε, σε κάποιους συγκεκριμένους ε, ομιλητές. Η κυρία που μίλησε για τη σχέση γεωργίας παραγωγής τροφίμων, ίσως είναι ερώτηση προς τον κύριο Ντρούγας, επίσης τα ερωτήματα προ τον κύριο Εγγενχόφερ ήταν ξεκάθαρα. Ε, κάποιος Πολωνός νομίζω έκανε κάποιε ερωτήσει που θα ήθελα να τι απαντήσει ο κύριο Γκενχόφερ, γιατί ε, τέθηκε, το πολύ σημαντικό ζήτημα των ιδίων πόρων. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω να υπάρξει εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δούμε όμω, ε, θα μα πει το πάνελ. Μετά ένα ρωμανικό ερώτημα νομίζω και να ρωτήσουμε τον κύριο Μπόλτ πώ μπορούμε να διδαχθούμε από τι χρηματοπιστωτικέ αγορέ για τι ενεργειακέ αγορέ και να έχουμε αυτή την αγοροκεντρική δομή. Θα ήθελα να μα ε, πείτε κάποια πράγματα περισσότερο πάνω σε αυτό. Και τέλο, ε, σχέση τροφίμων ενέργεια. Να κάνουμε μια σύνθεση και σύνοψη που θα μπορούσε δηλαδή ο καθένα να πει την άποψή του. Λοιπόν, κύριο Σίγκενχόφερ, πρώτο το λόγο. Uh, yeah, uh, yeah, there were a number of, of... Πράγματι υπήρξαν κάποια ζητήματα που αφορούσαν εμένα προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι είναι δήλωση αποστολή ε, η στρατηγική Ευρώπη 2020. Και νομίζω κάπως παρεξηγήθηκε κάτι που είπα. Ε, είναι σημαντική η δήλωση αυτή, αλλά δεν θα πρέπει να την συγχαίουμε και ούτε να είμαστε κάπως υπερβολικά ακτιβιστές και να έχουμε και όλα αυτά που είδαμε στη στρατική της Λισαβόνας. Λοιπόν, ηγεσία, διαφορετικές τεχνολογίες. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Κίνα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα και εμείς είμαστε σχετικά μικροί σε σύγκριση. Φυσικά και η νεζική αγορά θα είναι ε, πάντοτε μεγαλύτερη αφού έχει τριπλάσιο πληθυσμό και αυξάνει το ΑΕΠ πάρα πολύ γρήγορα στη χώρα αυτή. Τι θα πει λοιπόν αν η Κίνα είναι ηγέτης ε, στην αιωλική ενέργεια παραδείγματος χάρη γιατί έχουν περισσότερες ανεμογεννήτριες ε, ή παρέχουν τεχνολογία. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρα. Αυτό το ζήτημα με τους αριθμούς, με τα νούμερα Πρόσφατα δημοσιεύσαμε ένα βιβλίο για ε, θέματα που αφορούν το κλίμα και εκεί είναι ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο ότι οι εκπομπές του του άνθρακα της Κίνας σε εξαγωγές τους είναι πενταπλάσιες σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Σας προσέχουμε λοιπόν κινέζικη αποδοτικότητα, αλλά πάνω ε, πενταπλάσιες εκπομπές του του άνθρακα και το ίδιο ισχύει και για την Ινδία. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για αποδοτικότητα, περιβαλλοντική απόδοση των χωρών αυτών. Διαλέξτε όποιον δείκτη θέλετε. Μπορεί να είναι λίγο παραπλανητικός όμως. θέλαμε παγκόσμια συμφωνία για απόλυτα όρια στις κλιματικές αλλαγές και τώρα περνάμε σε μια άλλη ε, αντιμετώπιση και σε μια άλλη προσέγγιση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ηγέτης όλες τις τεχνολογίες. Μπορούμε να είμαστε ε, πρωτοπόροι σε κάποιες τεχνολογίες, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είμαι σε όλα. Παραδείγματος χάρη, αιωλική ενέργεια, ε, ηλιακή συγγνώμη, ενέργεια. Έχουμε τους ηλιακούς ε, συλλέκτες. Γιατί θα πρέπει η Ευρώπη να προσπαθεί να πάρει ταινία σε όλες τις αγορές. Ε, μπορεί να χάσουμε εκεί. Ή ανεμογεννήτριες πώς μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από την Κίνα στην Ευρώπη. Υπάρχουν ολοκληρωμένες διαδικασίες και ίσως εκεί πράγματι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε πρωτοπόροι σε όλα. Όχι. Επίσης, πάλι δεν ξέρω αν με καταλάβατε εντελώ, είπα ότι πράγματι ε, η κατεύθυνση του προπολογισμού, η προβασικός προσανατολισμό πρέπει να είναι ξεκάθαρος, γιατί αλλιώ μπορεί να υπάρξουν ε, προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διάθεση των κονδυλίων. Τα κίνητρα πρέπει να είναι σωστά ακόμη και για πιο φτωχές οικονομίες, για να περάσουν δηλαδή προς μια τεχνολογία χαμηλή σε διοξίδιο του άνθρακα. Και αυτό να μην το κάνουν μόνο οι πλούσιες χώρες που μπορούν να το κάνουν από οικονομικής πλευράς και όπου έχουν και την απαραίτητη τεχνολογία. Δεν λέω ότι το χρήμα δεν είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει πολιτική καθοδήγηση και μετά θα δούμε. Μετά μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Η κοινοτική τώρα πτυχή της ε, ενωσιακής χρηματοδότησης και πάλι θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Στο σκέλος της συνοχής, φυσικά και είναι σαφές ότι μιλάμε για ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκές δαπάνες, αλλά η αριστεία, έρευνα και ανάπτυξη, υψηλή τεχνολογία, high tech, ε, ο Σάπη νομίζω το ανέφερε, η ηγεσία εδώ βρίσκεται σε κάποια από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη και θα πρέπει να το δεχθούμε να μην είμαστε υπεραισιόδοξοι για την προστιθέμενη αξία για κάποιες από τις μεγάλες χώρες με τις πολύ σημαντικές τεχνολογικές δυνατότητες. Επίσης, ήδη οι πόροι, ETS, το σύστημα αυτό ανταλλαγή ε, δικαιωμάτων εμπορία και αν μπορεί να είναι ίδιο πόρο. Ε, το σκεφτόμουν και μάλιστα το Μάρτιο του 2008 έχει δημοσιευθεί και μια έκθεση. Είναι διαθέσιμη η έκθεση αυτή. Και είναι σαφέ ότι αν μιλάμε για ένα νέο πόρο, αυτό μπορούσε να είναι ο πρώτο που θα σκεφτόταν κανεί, διότι πληρεί όλα τα κριτήρια ενό ευρωπαϊκού εσόδου. Εδώ βέβαια θα ακολουθήσω τη γραμμή του Αντρέ Σαπίρ. Εμεί κάναμε την ανάλυση και εσείς ως πολιτικοί θα πρέπει να λάβετε την απόφαση. Φοβούμε ότι η απόφαση αυτή δεν είναι καν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Ευρωκοινοβουλίου. Βέβαια, μακροπρόθεσμα θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή την αρμοδιότητα, αλλά μάλλον είναι δύσκολη προς το παρόν η μάχη που θα πρέπει να δοθεί και δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Pierwsza kwestia dotycząca pewnej autarki energetycznej. Η πρώτη παρατήρηση αφορά την αγορά της ενέργειας. Έχουμε τεχνολογίες τις οποίες γνωρίζουμε σήμερα, αλλά δεν πάβουν να είναι ακριβές. Κάτι το οποίο τις εμποδίζει να γίνουν πιο εκδημοκρατισμένες με την έννοια ότι να έχουν μεγαλύτερη διάδοση. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε όπως σας είπα, να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα μέσα μέσω ενός κοινού προϋπολογισμού και το σύνολο αυτών των ε, μέσων να είναι διαθέσιμα πολύ περισσότερο από σήμερα. Οι πρώτες ύλε, οι οποίες παράγονται ε, στον τομέα της γεωργίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει αντικείμενο μεγαλύτερης ενασχόλησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από αρκετά χρόνια ο τομέας, σαν παράδειγμα των τιμών των τροφίμων, ήταν σχετικά ελεγχόμενος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια με τις τεχνολογικές εξελίξεις, με τις τελεπικοινωνίες, με την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, Όλα τα άλλαξαν και φυσικά άλλαξε και η αγορά των τροφίμων. Και ήρθαν εδώ και πάρα πολλοί κερδοσκόποι όπως και σε πολλές άλλες αγορές. Οι παγκόσμιες αγορές τα τρόφιμα έχουν πλέον αλλοιωθεί και ένα άλλο θέμα το οποίο συνδέεται με αυτό είναι οι ανανιώσιμες πηγές ενέργειας που βασίζονται στις πρώτες ύλες. Αν οι πρώτες είναι ακριβές, τότε αποκλείουμε κάποιες μορφές ενέργειας τέτοιου είδους. Αν όμως το κόστος είναι ελεγχόμενο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και οι γεωργοί και αυτοί ακολουθούν. Υπάρχει επίσης και ένα θέμα εδώ νοοτροπίας θα έλεγα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι έχουν κάνει οι Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει μια βοήθεια για την παραγωγή πρώτης ύλης η οποία θα οδηγήσει στην παραγωγή ενέργειας γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα αποδοτικό οικονομικά. Θα πρέπει επίσης ε, να θυμόμαστε όλοι ότι το βασικό είναι ε, τα τρόφιμα σε σχέση με τη γεωργία. Βασικός μας στόχος είναι να θρέψουμε πρώτον την, ε, τον ευρωπαϊκό πληθυσμό φυσικά και να βοηθήσουμε στη διατροφή και του υπόλοιπου κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα η αγορά της ενέργειας είναι σε λειτουργία πραγματική. Ναι, φυσικά είναι. Νομίζω ότι αρκετά πράγματα έχουν προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι η αγορά φυσικού αερίου παρά το ότι όλη η παραγωγή φυσικού αερίου όπως οι ρωσικές, οι νορβηγικές κτλ πολεμούν για μακροπρόθεσμα προγράμματα, οι τιμές ε, κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Έχουμε μια τιμή σποτ για το φυσικό αέριο που είναι 30% χαμηλότερη από τις προβλέψεις της μακροπρόθεσμες και αυτό παρά την μαζική αντίσταση των ε, μεγάλων εταιριών. Δουλεύουν λοιπόν οι αγορές ενέργειας αλλά απαιτούνται περισσότερες μορφές ελέγχου, όχι ελέγχου, εποπτείας μάλλον, έτσι ώστε και μέσω των κατάλληλων νομοθετικών προτάσεων για την διακανονιστική εποπτεία των αγορών ενέργειας γιατί δεν ελέγχονται σωστά οι αγορές αυτές απαιτείται περαιτέρω διακανονιστική ρύθμιση αλλά θα πρέπει να γίνεται αυτό μέσα σε αγορές μεγάλες που να ξεπερνούν το μέγεθος μιας χώρας βέβαια, να έχουν περιφερειακή τουλάχιστον διάσταση, να είναι διαφανείς οι αγορές και έτσι θα δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα και για τους επενδυτές και για τους καταναλωτές έτσι ώστε αυτές οι αγορές να μην θεωρούνται ακριβές και να είναι ασφαλείς και μακροπρόθεσμα και δυνατότητες επιλογής να δίδονται από τη μία ενέργεια στην άλλη. Τι μπορεί να κάνει κανείς προς την κατεύθυνση αυτή, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί μέσα σε πέντε μόνο λεπτά. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου θα ήταν καλοδεχούμενες οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και όπου κανένας μπορεί να προχωρήσει με μια κάποια εμπιστοσύνη. Στον τομέα των ηλεκτρικών δικτύων απαιτείται διαρρύθμιση τέτοιου είδους έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης από εναλλακτικέ πηγές όπως η αιωλική ενέργεια, απαιτούνται περισσότερες δυνατότητες διασύνδεσης και εδώ απαιτούνται κάποιες επενδύσεις και απαιτούνται περίπου 20 με 30 δις κατέτος επιπλέον τα επόμενα 10 χρόνια και κάθε βοήθεια από την Ευρώπη είτε στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του 2020 είτε όχι είναι καλοδεχούμενη. Θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε και την παραγωγή ενέργειας εκτός καυσίμων. Αυτό ισχύει για την φωτοβολταϊκή ενέργεια και για την θερμική, γεωθερμική ενέργεια ότι δεν απαιτεί δηλαδή καύσιμα και ε, βοηθάει τα θέματα ε, τα οποία μας ενδιαφέρουν, δηλαδή τα γεωργικά προϊόντα. Και αν δει τελικά κανείς και την έκθεση για τη διεθνή ενέργεια που δημοσιεύτηκε πριν μερικές εβδομάδες, απαιτείται να έχουμε μια παραγωγή ηλεκτρισμού το 2050 συγγνώμη, ελεύθερη από εκπομπές καυσαερίων διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι πάρα πολύ φιλόδοξο και θα έλεγα ότι πηγαίνει προς την κατεύθυνση αυτή, ότι δηλαδή προείπα προηγουμένως είναι καλοδεχούμενο. Και τέλος, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης η Ευρώπη δίνει πάρα πολύ αιμονή ε, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει έρευνα και ανάπτυξη για τα φωτοβολταϊκά σαν παράδειγμα αλλά υπάρχουν πολλά μέρη της Ευρώπης που είναι κατά καλά οργανωμένα σε τεχνολογικό επίπεδο και πρέπει να φανούμε πιο φιλόδοξοι όπως οι έξυπνες πόλεις, όχι μόνο τα ηλεκτρικά συστήματα αλλά και τα συστήματα ηλεκτρικής αποτελεσματικότητας, να χρησιμοποιήσουμε το συνδυασμό των αποτελεσματικών τεχνολογιών στον τομέα της ηλεκτρονικής και εδώ έχουμε έναν τομέα ο οποίος δεν είναι εύκολος για άλλες χώρες όπως η, Μέση Ανατολή να μας προλάβει θα έλεγα, η Άπο Ανατολή συγγνώμη, γιατί εκεί υπάρχει μία απόσταση και μία θα έλεγα υστέρηση σε ορισμένου τομεί. Αν λοιπόν προσπαθήσει κανείς να χρησιμοποιήσει αυτά τα δίκτυα με έξυπνο τρόπο, μέσω ακριβώς του συστήματος των έξυπνων δικτύων, αποκτά κάτι περισσότερο από συγκριτικό πλεονέκτημα γιατί θα έχουμε την δυνατότητα χρήσης των φωτοβολταϊκών που μπορεί να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να κατασκευαστούν στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να έχουμε σαν στόχο την παραγωγή φθηνότερης φωτοβολταϊκής υποδομής από ότι εκτός Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι γενικά η παραγωγή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και σε οργανωτικό επίπεδο επίσης μπορούμε να κάνουμε πράγματα καλύτερα από άλλους και πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, ομιλητές, τους ομιλητές από την πλευρά της Επιτροπής σας. Δεν θέλω ε, να μακρηγορήσω, αλλά Κάναμε μια συζήτηση δυόμιση ωρών. Νομίζω ότι στην κοινή αυτή αγορά ε, μπορούμε να αναζητήσουμε πολλά. Όπως είπαν ε, οι τρεις ομιλητές του πάνελ, αν η Ευρώπη καταφέρει να συνδυάσει την ανάγκη για νέα δίκτυα, ε, την ανανεώσιμες πηγές, την αγοροκεντρική προσέγγιση, ίσως αργότερα ήδη οι και ένα σωστό αντιστάθμισμα μεταξύ βιοκαυσίμων και παραγωγής τροφίμων, και βελτιστοποιημένη και ολοκληρωμένη χρήση. Και γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί νομίζω ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες και αφορούν την καθημερινότητά τους, αφορούν τη θέρμανση των σπιτιών τους, ε, τη στέγασή τους, το τι τρώνε, πώς ζουν. Και όλα αυτά που διακυβεύονται σε επίπεδο παγκόσμιο, νομίζω ότι αν υποθούν με διαφορετική γλώσσα ε, θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Αν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδυάσει, νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ καλή κοινή αγορά ενέργειας. Ευχαριστώ και θα... Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το δεύτερο πάνελ. Νομίζω ότι πραγματικά τέτοιου είδους πάνελ λειτουργούν αρκετά καλά και παρουσιάζουν καινούργιες ιδέες, καινούργιες προσεγγίσεις. Πράγματι ο τίτλος τώρα της, του θέματός μας όπως παρουσιάζεται εδώ ε, έκρυβε πολλά μυστικά και Πραγματικά υπάρχουν, ε, παρόλο που ασχολούμεθα με όλα τα θέματα αυτά εδώ και πολύ καιρό, ε, υπάρχουν και εκπλήξεις. Ελπίζω τώρα ο εισηγητής να μ' ακούει, γιατί η δική του δουλειά είναι τώρα να κλείσει την πρώτη μέρα της ακρόασης να εξάγει τα συμπεράσματα της πρώτης μέρας και εγώ σας καλώ στις 6.30 ώρα στο τέλος αυτής της πρώτης μέρας της ακρόασης ε, σας καλώ να πιούμε ένα κοκτέιλ ο εισηγητής ο κύριος Γαρίγα Ευχαριστώ πολύ ήταν πάρα πολύ ψηλού επίπεδου οι ομιλητές στα δύο πάνελ. Ε, ήταν πολύ σημαντικά τα συμπεράσματα ε, στα οποία θα μπορούσα να καταλήξω, αλλά ακόμη δεν είναι προφανή για μένα, διότι κάθε ένας από τους εισηγητές ε, εξέφρασε ιδέες καινοτόμε, θα έλεγα, που πολλές φορές η μία αντιφάσκει ε, με, με τις κατευθύνσεις που είχα στο μυαλό μου για την εκπόνηση της έκθεσης. Τι θέλω να πω βέβαια με όλα αυτά, ότι ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η όλη συζήτηση, αλλά υπήρξαν και επίμαχα θέματα. Όλα αυτά που άκουσα, όλες τις απόψεις θα τις λάβω υπόψη και θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω τα σχετικά στα έγγραφα, στο έγγραφο εργασία στο οποίο εκπονώ. Τώρα, για να συνοψίσω τα δύο πάνελ ως εισηγητής ε, που θα πρέπει να εκπονήσω ένα έγγραφο εργασίας ε, προτού τοποθετηθεί συνολικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ε, προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές. Θέλω να πω ότι αφού άκουσα το πρώτο πάνελ, έχω περισσότερες ανησυχίες σε σχέση με πριν για το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 στις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικέ. Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια ευκαιρία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να αντιχάσει Εάν αποτύχει η στρατηγική 2020, είτε γιατί δεν συμμετέχουν επαρκώ τα κράτη-μέλη, είτε γιατί δεν είμαστε ικανοί να ορίσουμε έναν προϋπολογισμό που θα είναι επαρκής και προσδιορίσιμος ό,τι αφορά τους διάφορους στόχους στρατηγικής, αυτό θα ήταν μια σημαντική ευρωπαϊκή αποτυχία, ιδίως όταν μιλάμε για μια στρατηγική που όπως αναφέρατε και εσείς έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφή ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι ε, κάτι που δύσκολα μπορεί να συμπεριλάβει κανείς ε, στις μελλοντικές ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Η συζήτηση των εγγράφων προβληματισμού Δείχνει ότι ούτε και στην Επιτροπή Σούρε δεν υπάρχει ομοφωνία σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Αυτό το smart growth, η ευφυής ανάπτυξη θα πρέπει να είναι οριζόντιο που θα συμπεριλαμβάνει τα διάφορα κονδύλια που ήδη υπάρχουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό ή μήπως πρέπει να είναι ένας ξεχωριστός πυλώνας και ένας αυτοσκοπός στο πλαίσιο της ε, μελλοντικής μουσουλμικής προοπτικής. Φυσικά και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσουν ε, τα μέλη της Επιτροπής ΣΟΥΡ και νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια των μελών του πάνελ. Εξίσου ενδιαφέρον ήταν και το ζήτημα της έρευνας. Στο μέλλον, τι θα γίνει με την τάση αυτή που υπάρχει. Έχουμε την ε, συνοχή από τη μία πλευρά, την αριστεία από την άλλη και υπάρχει μια ένταση, αν θέλετε, μεταξύ αυτών των δύο. Πολιτική έρευνας, πολιτική ανταγωνιστικότητας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούνται πολιτικές αυτές ε, σε μεγάλο ποσοστό από την πολιτική συνοχή. Αυτό ισχύει για τις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά εάν θέλουμε να βρούμε μια διασύνδεση με έναν δεσμό μεταξύ των ολοντικών δημοσιονομικών προοπτικών και της στρατηγικής 2020, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ορίσουμε και ίσως ε, να διαχωρίσουμε ξεκάθαρα. Δηλαδή να πούμε σε ποιο βαθμό θα πρέπει να είναι η πολιτική συνοχή ανεξάρτητη από την πολιτική έρευνα και καινοτομία. σω, παραδείγματο χάρη, λαμβάνοντα υπόψη ότι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο μπορούσε, παραδείγματο χάρη, να, χρησιμο... να χρηματοδοτήσει τι περιφέρειες που μπορούν να είναι κέντρα αριστεία Και τα διαρθρωτικά ταμεία, όπω έχουν σήμερα ή όπω θα έχουν στο μέλλον, θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να επικεντρωθούν στι περιοχέ συνοχή. Δεν ξέρω, όλα αυτά ε, είναι ανησυχίες ε, που εξέφρασαν στην Επιτροπή μας τα μέλη του πάνελ. Υπάρχει πάντως ένα θέμα το οποίο υπάρχει ομοφωνία και, και σαφήνεια, δηλαδή ότι στις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να δοθεί ε, μεγάλη έμφαση στις εκπαιδευτικές ε, πολιτικές, στις πρωτοβουλίες για την καινοτομία, έρευνα, όλοι οι, οι ομιλητές το ένα δις ευρώ εκεί θα το επένδυαν. Όταν λοιπόν συμφωνούν όλοι αυτοί οι διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες ότι τα χρήματα θα πρέπει να μπουν σε ένα συγκεκριμένο κορβανά, μάλλον έχουν δίκιο. Θα τους προσέξουμε λοιπόν και θα λάβουμε υπόψη τις υποδείξεις τους. Εκπαίδευση, έρευνα, ανάπτυξη, όλοι αυτοί οι τομείς θα πρέπει να είναι επίκεντρο των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη βιωσιμότητα, το δεύτερο πάνελ, πράγματι θα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στον ενεργειακό τομέα και αυτό μας ανησυχεί γιατί μέρος των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών θα πρέπει να αντισταθμίσουν το σφάλμα το οποίο διαπράχθηκε στις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές ήτι δεν υπήρχαν επαρκείς πόροι για τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων εν γέννη και δι για την κατασκευή υποδομών ενεργειακών tens η Δεν είχαν τα δίκτυα αυτά σχεδόν, θα έλεγα, καμία χρηματοδότηση και αυτό θα πρέπει να αλλάξει στο μέλλον. Εξίσου ξεκάθαρο είναι ότι όλοι οι συγητές, όλοι, όλα τα μέλη του πάνελ τονίζουν ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να προσπαθήσει να ισοσταθμίσει τις ε, μελλοντικές υποδομές από ενεργειακής πλευράς και αυτή η συζήτηση ήδη γίνεται και για τα ευρωομόλογα που συζητάμε και για τις ε, συμπράξεις δημοσιοδικού τομέα και είναι προφανές ότι και η Επιτροπή ΣΟΥΡ θα προσπαθήσει να διερευνήσει τους μηχανισμούς αυτούς όπως τα δικαιώματα εμπορίας εκπομπών ε, ως μια νέα μέθοδο για την χρηματοδότηση των ενεργειακών δικτύων. Είπε ένα συνάδελφο ότι θα πρέπει να μπει ε, στο τραπέζι, να τεθεί επιτάψη αυτό το θέμα. Και σε σχέση και εν ώψη του 2015 επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη αυτή τη στρατηγική. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, ε, βιώσιμη ανάπτυξη, είναι σαφές ότι είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την αναθεώρηση της γεωργική πολιτική, όπω ξεκίνησε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τους στόχους που έχει, δηλαδή και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και σε ό,τι αφορά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα. Τέλος, ένα εργαλείο της δημοσιονομικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα κίνητρα. Τα κίνητρα προς ε, μια γεωργία και προς μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμες, ε, και θα πρέπει να δούμε και τη σχέση κόστους-οφέλους όταν θα χρηματοδοτήσουμε και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και τον γεωργικό τομέα που εξακολουθούν για μας να αποτελούν κλειδί για το μέλλον στο πλαίσιο των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών. Δεν μας ε, διαφωτίσατε γιατί αυτό είναι αποστολή των πολιτικών σε ό,τι αφορά την κατανομή των πόρων και τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σε όλους αυτούς τους τομείς, ε, τουλάχιστον μας ε, ε, γύρατε, θα έλεγα, νέε ανησυχίε και νέε αμφιβολίε που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες για τη δημιουργική άσκηση στην οποία θα πρέπει να προβούμε. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και πραγματικά πετύχατε το στόχο σας οι ομιλητές ε, μιλώντας σε εμάς πολιτικούς. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μέρας είδαμε ότι διαπιστώσαμε ότι με τη στρατηγική της Λισαβόνας δεν επιτύχαμε τους στόχους μας. Είμαστε αισιόδοξοι σε σχέση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, αλλά ένα πράγμα είναι ήδη σαφές. Αν δεν αποφασίσουμε από κοινού τα σωστά μέτρα, αν για να εφαρμόσουμε τελικά την στρατηγική Ευρώπη 2020, αν δεν καταρτήσουμε το σωστό προϋπολογισμό για τις αλλαγές αυτές, τότε φταίει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, ελάτε να πιούμε ένα ποτήρι.